όπως ε, βλέπετε είναι πολύ ενδιαφέροντα τα θέματα και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να περάσουμε στην έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Και... Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Και τώρα έχω την τιμή να σας ε, καλωσορίσω σε ένα πολύ βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η αποστολή επιτήρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχέση με τη Γεωργία, αποκλειστικά με τη Γεωργία. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να ε, τηρήσω το πρωτόκολλο, να καλωσορίσω την κυρία Πρέσβη, εκπρόσωπο της ε, Γεωργίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Ναταλή Σαμπανάτζε. Την ξέρουμε την κυρία Σαμπανάτζε, έχει έρθει πολλές φορές στην Επιτροπή μας και την καλωσορίζουμε. Εξ αριστερών μου κάθεται ο κύριος Κένεθ Ντίν, Διευθυντής της Μη Στρατιωτικής Δυνατότητας Σχεδιασμού και Διεξαγωγής Επιχειρήσεων. Και επίσης έχουμε έναν εξίσου ε, σημαντικό ομιλητή, αρχηγό της Αποστολής Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία, τον κύριο Κεστούτης Γιανκάουσκας. Ε, τον έχω γνωρίσει ε, όταν ε, τον επισκέφτηκα επί τόπου στην έδρα του, αλλά βεβαίως είναι η δική του πρώτη επίσκεψη εδώ. Τους καλωσορίζουμε όλους και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον κύριο Κένετ Ντίν και μετά στον κύριο Κεστούτης Γιανκάουσκας και κυρία Σαμπανάτζε. Θα δώσω το λόγο σε εσά για να ολοκληρώσουμε με εσά τη συζήτηση για να μας δώσετε έτσι μια γενική εικόνα της ε, ασφάλειας, των θεμάτων ασφαλείας ε, σε σχέση με τη Γεωργία. Κύριε Ντίν, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρέσβη, αγαπητοί ε, Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Για μένα, ως επικεφαλής, ως αρχηγός της αποστολής, είναι μεγάλη τιμή το ότι βρίσκομαι εδώ σήμερα σε εσά. Επίσης, χαίρομαι πάρα πολύ που ε, έχουμε και τον κύριο Γιανκάουσκας που δεν είναι μόνο αρχηγός της επιστολής, ε, της αποστολής επιτηρής, αλλά είναι επίσης και ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης, ε, τον οποίο λυσεύονται, έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Έτσι δηλαδή μπορούμε να είμαστε ησυχοί ότι η αποστολή αυτή βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Η αποστολή στη Γεωργία είναι μία από τις αποστολές με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι ένα σημαντικό κομμάτι της συμφωνίας που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποστολή εξακολουθεί να ε, διεκδικεί ένα στόχο που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να υπάρχει ε, ειρηνευτική αποστολή επιτόπου. Από το 2009 αυτή η επιστολή είναι η μόνη παρουσία διεθνών δυνάμεων στη Γεωργία. είναι καθοριστικός παράγων για τη σταθερότητα στη Γεωργία και γενικότερα για την περιοχή της Μεσογείου. Και νομίζω ότι αυτό το δέχονται τα περισσότερα από τα εμπλεκόμενα μέρη και στη Γεωργία και εκτός αυτής η αποστολή ε, διαδραματίζει ένα καθοριστικό στοιχείο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να φέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η αποστολή αυτή αποφέρει ωφέλεια αλλά και είναι και μια θετική παρουσία ε, στη Γεωργία και γνωρίζω πολύ καλά ότι μετά θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Θα θυμάστε ότι τον Ιούλιο του περασμένου έτους ε, υπήρξε κλιμάκωση της ένταση, η οποία μεταξύ άλλων προκλήθηκε και από την εγκατάσταση ε, ε, καθοριστικών γραμμών στα σύνορα. Σήμερα υπάρχει επιτόπου υπάρχουν ένοπλες δυνάμεις, ε, κυρίως εκεί που ε, ορίστηκαν τα σύνορα και ως εκ τούτου προέκυψε κλιμάκωση της έντασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε πάρα αυτά και νομίζω ότι έστειλε την αποστολή στις 24 Σεβδόμου αλλά επίσης ε, και δρομολογώντας ένα διάλογο ε, με ε, αναφορές σε πραγματικό χρόνο. Αυτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να μην επεκταθεί και κλιμακωθεί περαιτέρω η βία και η ένταση, να μην παραταθεί η κατάσταση. Η αποστολή λοιπόν είναι καθοριστική σημασίας. Βεβαίως το θέμα δεν είναι ότι αφορά μόνο τα σύνορα, αλλά αφορά και όλα αυτά που είναι τα συνεπακόλουθα της ε, ε, ειρηνευτικής διαδικασίας, το τι διαδραματίζεται σε αυτά τα σύνορα. Από τη μία και από την άλλη πλευρά. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί την κατάσταση και να προσπαθεί να καθησυχάσει όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Να σας πω ότι όσον αφορά αυτή την αποστολή στη Γεωργία, για μας ε, είναι ένα κράτος με το οποίο θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις, αλλά αυτό που έχει σημασία από επιχειρησιακής πλευράς είναι ότι ε, εκεί επιθυμούμε να υπάρχουν ε, εκπρόσωποι μας με πραγματικές ε, ουσιαστικές ικανότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτή την εισαγωγή και σας δίνω και πάλι το λόγο. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο και στούτη Γιάν Κάσκα, αρχηγό τη Αποστολή Επιτήρηση Ευρωπαϊκή Επιστροπή στη Γεωργία. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ε, τιμή για μένα να είμαι εδώ ενώπιον σα σήμερα έτσι ώστε να σας παρουσιάσω την εργασία της Επιτροπής Επιτήρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Ε, και μάλιστα είχα τη χαρά ε, να έχω μερικούς από εσά ε, στην Τυφλίδα και πραγματικά αυτές οι επισκέψεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να έρχεστε Και Θα ήθελα να σας παρουσιάσω στο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εργασία. Να σας ευχαριστήσω για την εργασία που κάνετε εσείς εδώ καθώς επίσης και η CCPC επιτόπου. Είναι πάρα πολύ ε, ευρεία η αποστολή μας, όχι μονάχα για τη Γεωργία, αλλά και για τον ε, Νότιο Κάφκασο. Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι στην ε, σταθερότητα και την ειρήνη της περιοχής και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσει και η πρέσβης της Γεωργίας μετά από λίγο. Το 2008 ξεκινήσαμε την αποστολή μετά από διάφορες εχθροπραξίες που έλαβαν χώρα εκεί και συνεχίζουμε την επιτήρηση. Από το 2009 ε, η ε, αποστολή μας είναι η μοναδική σημαντική διεθνής παρουσία επιτόπου. Ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ήδη κάνει περίπου 50.000 περιπολίες και έχουμε παρουσιάσει πολλές ενημερώσεις και εκθέσεις. Επίσης, το περισσότερο προσωπικό μας είναι στα πλαίσια των διοικητικών συνοριοκών γραμμών, δηλαδή την Administrative Boundary Line ε, και πρέπει να σας πω ότι παραμένουμε επιτόπου ε, ε, διότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να παραβιάζει το σημείο 5 των, των 6 σημείων της συμφωνίας που είχαμε κάνει. Έχουμε επίσης, πρέπει να σας πω ότι είμαστε τα αυτιά και τα μάτια της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου. Έχουμε τρεις αξιωματικούς πεδίου κοντά στην διοικητική ε, γραμμή και ε, πάντα τίνουμε βίκο νούσε εις ε, αιτήματα του τοπικού πληθυσμού. Προσπαθούμε να λύσουμε παρεξηγήσεις και να δώσουμε αξιόπιστες πληροφορίες. Ορισμένοι μπορεί να σκεφτούν ότι τα 7 αυτά χρόνια είναι πάρα πολύ μακρά περίοδος για μια τέτοια επιτροπή. Θα ήμουν ο πρώτος που θα χαιρόταν εάν καταφέρναμε να φύγουμε σήμερα ή αύριο. Τα πράγματα προχωρούν αλλά δυστυχώς ακόμα δεν ε, έχουμε ε, φτάσει στο σημείο που θέλουμε γιατί η επούλωση των πληγών των πολέμων ε, είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Οι προσπάθειες για εξέβρεση βιώσιμης λύσης εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα και πιστεύω ότι εντωμεταξύ θα πρέπει να υπάρχει μια παρουσία σαν τη δική μας. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τις, τους εκπροσώπους της ε, ενωσιακής οικογένειας επιτόπου, δηλαδή την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης ε, και τον ειδικό εκπρόσωπο για τον Νότιο Κάφκασο. Ε, σε γενικές γραμμές, παρότι η κατάσταση είναι ήρεμη, παραμένει πάρα πολύ εύθραυστη και ακόμα δεν έχει καθόλου σταθεροποιηθεί. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από τα, τις καταστάσεις οποίες μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε και οι οποίες ενδεχομένως μπορεί να έχουν ε, σημαντικές ε, ε, επιπτώσεις. Θα θυμάστε ενδεχομένως τις ξαφνικές εντάσεις στα πλαίσια των, ή στη γραμμή των διοικητικών, της διοικητικής νοριακής γραμμής το προηγούμενο καλοκαίρι. Ε, ε, αυτές έλαβαν χώρα σε ε, χωριά τα οποία δεν ήταν πολύ γνωστά, τα Τσιτελουμπάνη και Ορκοσάνη. Αυτές οι εντάσεις ξεκίνησαν όταν οι de facto αρχές της Νότιας Οσετίας και της Ρωσικής Ασφάλειας έβαλαν κάποια περιοριστικά έτσι ώστε να δείξουν ότι εκεί σταματούν τα, τα σύνορα. Ε, αυτά ε, τα, τα, σήματα ε, είχαν, τα, είχαν εγκαταστήσει πολύ κοντά στην, στο, οδό η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική λόγω του αγωγού Μπακού Σούψα. Εμείς βοηθήσαμε έτσι ώστε οι ντόπιοι πληθυσμοί να έχουν πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο και να μην κοπούν οι δικές τους επαφές. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε επιτόπου παρόντες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την ε, εβδομάδα. Ε, ε, έχουμε επίσης, κάνουμε, καταβάλουμε επίσης προσπάθειες έτσι ώστε να φέρουμε σε επαφή όλους τους επιτόπου φορείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε μια αποδεκτή κοινά λύση. Ε, τέτοιου είδους ε, όμως ε, εντάσεις καταδεικνύουν την ανάγκη εξακολούθηση της παρουσίας της αποστολής επιτόπου. Φανταστείτε ε, εάν ε, ε, αυτού του είδους οι καταστάσεις και η εγκατάσταση τέτοιων hot spots συνέχιζε και για το μέλλον. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ ο ίδιος έχω συμμετάσχει σε περιπολίες και αποτελούν αυτές οι περιπολίες μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιου πληθυσμούς. Ε, το, το προηγούμενα χρόνια κυρίως, δεν το προηγούμενο ε, καλοκαίρι, ε, εμείς μπορέσαμε να μετρήσουμε τις, την παρουσία των ενόπλων δυνάμεων και είναι γεγονός ότι ορισμένες από τις στρατιωτικές βάσεις, κυρίως στην Απχαζία, είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και δημιουργούν προβλήματα προβλήματα ε, στους ντόπιου πληθυσμούς. Ε, επαγρυπνούμε ε, διότι η νέα σειρά στρατιωτικών ασκήσεων θα λάβει χώρα φέτος και επομένως ε, μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε. Η ελευθερία κίνησης επίσης είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και το παρακολουθούμε ε, από κοντά. Οι οικογενειακοί δεσμοί μερικές φορές απειλούνται. Ε, πρέπει να μπορούν οι κάτοικοι να πηγαίνουν ας πούμε σε κηδείες που, βρίσκονται, που γίνονται στην άλλη πλευρά ή να μπορούν να επισκέπτονται τα οικογενειακά κημητήρια. Έχουμε επίσης ε, πολύ συχνά κρατήσεις ε, ε, ατόμων, περιορισμό της προσωπικής τους ελευθερίας κλπ. Ε, τα σημεία περάσματος των πολιτών ε, είναι εξοπλισμένα με πάρα πολύ εξεζητημένα ε, συστήματα και αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στους πληθυσμούς. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περνούν καθημερινά αυτά τα σημεία ελέγχου, όπως παιδιά για να πάνε στο σχολείο ας πούμε. Ε, σας είπα ότι ε, εμείς είμαστε παρόντες 24 ώρες 24 ώρο ε, κάθε μέρα της ε, εβδομάδας και έχουμε και παρακολουθούμε ε, κυρίως ε, τις ε, καταστάσεις, όλες τις ασκήσεις, τις στρατιωτικές, οποιαδήποτε περίπτωση πυροβολισμού διαπιστώσουμε. Δουλεύουμε πάρα πολύ στην πλευρά της πρόληψης των ε, ε, εντάσεων σε συνεργασία με τον ε, τοπικό πληθυσμό. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί με, την, με τους εκπροσώπους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όλες ε, τις, ε, όλες τις προβληματικές καταστάσεις από αγνοούμενους μέχρι ε, κρατούμενους, φυλακισμένους και Και σε πολλές περιπτώσεις καταφέρνουμε να λύσουμε καταστάσεις. Βεβαίως ορισμένες ιδιαίτερως πολιτικές περιπτώσεις αναφέρονται στην Γενέβη. Στα πλαίσια δε της συνεργασίας μας με την Γενέβη κάνουμε μία αναφορά τέσσερις φορές ε, την εβδομάδα, ε, συγγνώμη το χρόνο, ε, στα πλαίσια της ομάδας εργασίας 1. Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Επιτήρησης ε, προσαρμόζεται στις ε, καταστάσεις ε, που βρίσκει επιτόπου. Πέρσι είχαμε ξεκινήσει την λεγόμενη διαδικασία βελτιστοποίησης και οι προσπάθειές μας έχουν δώσει καλά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να βρούμε τεχνικές λύσεις βελτιστοποίησης. Ε, και ε, ευελπιστούμε ότι η συνοριοποίηση θα συνεχιστεί, ίσως με λιγότερο έντονο ε, ρυθμό. Επίσης, σύντομα θα δημιουργηθούν και άλλα hot spots. Απλώς χρειάζεται δηλαδή να εγκαταστήσουμε περισσότερα σημεία ελέγχου. Εξακολουθεί να υπάρχει ε, ένα πρόβλημα ε, ασάφειας όσον αφορά τα, τα, έγγραφα τα οποία θα πρέπει να έχουν ε, αυτοί που περνούν τις γραμμές ελέγχου. Στην Αφχαζία έγινα κάποιε κάποιες νέες αποφάσεις οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύσουν από την 1η Απριλίου και που ενδεχομένως θα δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Επίσης ε, προχωρούμε την ε, λεγόμενη συνθήκη για την, ε, για την συμφωνία και την στρατηγική εταιρική σχέση με την Απχαζία, τρίτη Alliance and Strategic Partnership with Abkhazia. Ε, λαμβάνουμε ε, υπόψη σε αυτήν την συμφωνία, σε αυτό το σύμφωνο ε, και έναν αριθμό υποσυμφωνιών, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη υπογραφεί. Ποιες είναι τώρα οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Η κύρια πρόκληση κατά την άποψή μου είναι η έλλειψη πρόσβαση στην Απχαζία και την Νότια Οσετία. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται και να, λάβουμε όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το θέμα αυτό αυτό. Προσπαθούμε ε, ε, να συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε έτσι ώστε να βελτιωθεί ε, αυτή η πρόσβαση. Επίσης, η επαναενεργοποίηση της γάλι IRPM και των συνεδριάσεών της που σταμάτησε το 2012 είναι μια άλλη πρόκληση είναι πάρα πολύ απαραίτητος ο μηχανισμός αυτός έτσι ώστε να συνεχιστεί ε, ο διάλογος. Επομένως ευελπιστούμε και ξέρω ότι ε, πολλές ε, προσπάθειες γίνονται και καταβάλλονται σε διεθνές επίπεδο έτσι ώστε να ξαναρχίσει ο διάλογος αυτός. Επίσης υπάρχουν και κάποιες ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις όπως ας πούμε η πίεση της Γεωργίας ε, για μεγαλύτερη ευρωατλαντική ολοκλήρωση και ενδεχομένως κάποια απάντηση σε αυτήν την ε, προσπάθεια ε, οι κοινοβουλευτικές εκλογές τον, το φθινόπωρο του 2016 κάποιες γενικότερες ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Ουκρανία, τη Συρία και την Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Όλες αυτές είναι κινήσεις οι οποίες ενδεχομένως θα έχουν επίπτωση επιτόπου. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, ασάφεια ε, και την ε, αστάθεια οπωσδήποτε είναι σαφές ότι η Επιτροπή Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να παραμείνει επιτόπου. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε για την στήριξή σας και για μία ακόμα φορά θα ήθελα ε, να σας ε, ε, προσκαλέσω να έρθετε στην Γεωργία. Η διαδικασία είναι ανοιχτή, τα πράγματα ακόμα είναι ασαφή και επομένως υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαιη ότι οι συνάδελφοί μου θα θελήσουν να έχουν μαζί σας ε, μια ανταλλαγή απόψεων στη συνέχεια. Να σας ενημερώσω ότι οι συντονιστές της Επιτροπής μας ε, αποφάσισαν να σταλεί αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ε, στη Γεωργία στα τέλη Μαΐου. Στην τυρκουάζ εβδομάδα του Μαΐου. Τότε λοιπόν θα επισκεφθούμε τη Γεωργία και ελπίζω στην συμμετοχή των συναδέλφων στην αντιπροσωπεία αυτή. Να δώσω τώρα το λόγο στην αυτή σε εξοχότητα κύρια Ναταλή Σαμπανάτζε, πρέσβυρα της Γεωργίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι εδώ μαζί σας. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως προσωπικά για την υποστήριξη και που μου δίνετε το λόγο βέβαια και που έχετε δώσει και το λόγο σε εκπροσώπους από τη Γεωργία να μιλήσουν ενώπιον της Επιτροπής σας. Είναι ε, δυστυχώς ε, τα θέματα της ασφάλειας κάτι που δεν μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο. Για πολλούς λόγους βρίσκομαι εδώ. Πρώτα απ' όλα για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη τη δική μου προσωπικά αλλά και της κυβέρνησής μου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την αποστολή επιτήρησης, η σημασία της οποίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί για την ασφάλεια της χώρας μου. Θα ήθελα επίσης ε, να εκφράσω την εκτίμησή μου για το έργο ε, του αρχηγού της αποστολής επιτήρησης του κυρίου Γιανκάουσκας που είναι παρόν σήμερα, ο οποίος έχει ηγηθεί με πολύ αποτελεσματικό τρόπο της αποστολής ε, διατηρώντας την αμεροληψία της, ε, την αντικειμενικότητά της και τυχαίνει ε, της μέγιστης εκτίμησης στο έργο του. Επίσης, για μια ακόμη φορά δράτω με της ευκαιρίας για να σας υπενθυμίσω τη σημασία αυτής της ε, αποστολής, διότι οι επιπτώσεις της ξεπερνούν την ίδια τη γεωργία, όπως έχει σήμερα η κατάσταση, με όλο και μεγαλύτερους κινδύνους ασφάλειας στη γειτονιά της Ευρώπης, ανατολικά και νότια. Σίγουρα τέτοιες αποστολές είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να έχει έναν ρόλο πρωταγωνιστικό στα παγκόσμια δρόμενα. Επίσης, ε, η απόφαση ελήφθη πάρα πολύ γρήγορα από ε, το Συμβουλίο μετά τον πόλεμο του 2008. Υπάρχει λοιπόν ε, μια αποστολή 200 ατόμων που σε χρόνο ρεκόρ αναπτύχθηκε επιτόπου. Υπήρξε τεράστια υποστήριξη ε, της Ένωσης στη Γεωργία και αυτό δείχνει πόσο ε, δεσμευμένη είναι στην ασφάλεια και σταθερότητα για την περιοχή. παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αποστολή επιτήρησης, ο ρόλος της ως ένα πρωταγωνιστής ε, ασφαλείας ήταν πολύ σημαντικός. Εκτιμά η κυβέρνηση της Γεωργίας την ταχύτητα την ανταπόκρισή σας στην κρίση του 8 και στην σταθεροποίηση που επαναλαμβάνω ότι σε αυτήν συνεισφέρει τα μάλλα και η αποστολή. Τώρα, η αποστολή επιτήρησης ε, και η μη στρατιωτική δυνατότητα σχεδιασμού είναι πολύ σημαντικές, έχουν σαφείς εντολές και έχουν τη δυνατότητα να επιτήρουν και να επαληθεύουν τα γεγονότα, τα πραγματικά περιστατικά και βλέπουμε ότι ναι υπάρχουν πράγματα τα οποία λαμβάνουν χώρα. Υπάρχει ε, στρατιωτικοποίηση, απομόνωση της Αψχασίας και της Νότιας Συνεχίζονται αυτές οι επιχειρήσεις. Οι ρωσικές δυνάμεις ε, δημιουργούν φυσικά σύνορα ε, στις γραμμές κατοχής και αυτό θα επηρεάσει και το πώς θα παραμείνει ο πληθυσμός εκεί, αλλά ελαχιστοποιούνται και οι επαφές μεταξύ ε, των κατοίκων αυτών των ε, περιοχών και περιοριζονται τα δυνητικά ωφέλη από μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν για τη βελτίωση της ε, κατάστασης του πληθυσμού και για την εξέβριση τελικά και μια λύσης μετά από διαπραγματεύσεις σε αυτή τη σύγκρουση. Τώρα υπάρχουν δυνάμεις σε απόσταση με τα πόδια από την, μια βασική οδική αρτηρία στη Ρωσία είναι ευάλωτη η χώρα μας, επομένως, σε ξένες εισβολές θα έλεγα. Κατά βάση αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι η Γεωργία προσπαθεί να συνεχίσει την ζωή της ε, και να φέρει σε πέρα στις βασικές της προτεραιότητες. Δεν θα υπερβάλλω να πω ότι η παρουσία ε, της αποστολής ε, βοήθησε τη Γεωργία να συνεχίσει να το ευρωπαϊκό θεματολόγιο. Δεν θέλουμε να ανταποκρινόμαστε σε προκλήσεις και δεν θέλουμε να οξύνουμε ε, το έλλειμμα που ήδη παρατηρούμε στην ασφάλεια της περιοχής. Και η ε, εντολή της αποστολής είναι ακριβώς να μειώσει τις εχθροπραξίες, ε, την όξυνση και να συνεισφέρει στην σταθερότητα. Και έχει πετύχει πολλά, παρά το ότι δεν μπορεί να πετύχει εντελώς ε, την εντολή. Είναι ο μόνος διεθνής μηχανισμός που μπορεί αποτελεσματικά να αντιδρά σε συμβάντα που δυνητικά μπορούν να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση όπως παράνομες προσαγωγές κρατήσεις, ε, πυροβολισμοί, απαγωγές κτλ. Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Πάντα υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν επίσης με τη διέλευση αυτών των διοικητικών συνοριακών γραμμών. Άκρος πολύπλοκη διαδικασία που ε, δυστυχώς ε, βλέπουμε να υπάρχουν πολλές καταχρήσεις. Η αποστολή διευκολύνει την πρόληψη και ανταπόκριση στα συμβάντα, το σχετικό μηχανισμό. Είπαμε για αυτή την ε, hotline, είναι πολύ σημαντική αυτή η γραμμή. Απ' την άλλη πλευρά, τα IPRM στην Αυγαζία δυστυχώς δεν έχει ε, ακόμη ε, επιτύχει τους στόχους της. Επίσης υπάρχει συμμετοχή στις διεθνείς συνομιλίες της Γενέβης με στόχο την εξέβρεση λύσης σε υψηλό επίπεδο. Η αποστολή ε, παρέχει πληροφορίες αντικειμενικές, αμερόληπτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην όλη διαδικασία, που είναι σημαντική η διαδικασία. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα οδηγήσει σε γρήγορη διευθέτηση του πρόβληματος, πάντως ε, μειώνει τους πολιτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ασφαλείας. Οι συνομιλίες της Γενέβης βλέπουν τι γίνεται με την κατάσταση ασφαλείας και στην και στην Απχαζία και αντιμετωπίζουν τα πιο επίγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα. Στον αφορά τώρα την τελική διευθέτηση. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που θα επηρεάσουν τα πράγματα, ιδίως τα γεωπολιτικά συμφέροντα διαφόρων παραγόντων για να μην πω ιδίω ενό. Μια από τι σημαντικότερε προκλήσει για την αποστολή, το είπατε, είναι η έλλειψη πρόσβαση στι κατεχόμενε περιοχές. Ελπίζουμε να αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Ταυτόχρονα όμω, αυτό αποτελεί πενθύμηση προ την Ένωση και τη διεθνή κοινότητα ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει τη Συμφωνία Κατάπαυση του Πύρος του 8, για την οποία διαμεσολάβησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εκεχηρία δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το όλο πλαίσιο και την κατάσταση ασφαλείας στη γειτονική, στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκαν τα σχετικά και θέλω να το τονίσω κι εγώ. Η αποστολή επιτήρησης είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που έχουμε για την ασφάλεια στην περιοχή. Η πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί την ασφάλεια προτεραιότητα έναν από του τομεί όπου θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερα μέσα και μηχανισμοί, έτσι έχει διακηρύξει και ένα πολύ καλό τέτοιο παράδειγμα είναι η αποστολή επιτήρηση. Ε, ιδίω όταν αυξάνονται κίνδυνοι για την ασφάλεια, είναι γνωστά αυτά, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε εδώ. Νομίζω ότι τέτοιε αποστολέ πρέπει να ενισχυθούν έτσι περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω ότι η συνεδρίασή μας ε, γίνεται σε συνεδρίαση με σε συνδυασμό με τις αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γεωργίας, Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν που λαμβάνουν και αυτές χώρα. Είναι λοιπόν χαρά μου το ότι μπορώ να καλωσορίσω τον κύριο Σέτσεκ Καλίμ, ε, ο οποίος είναι πρόεδρος αυτής της αντιπροσωπείας. Κύριε Καλίμ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω όλους. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συμμετέχω κι εγώ στην ανταλλαγή των απόψεων. Νομίζω ότι μπορώ να σας εκφράσω και τη δική μου την προσωπική άποψη με την έννοια ότι είδα επιτόπου την ε, πολύ σημαντική δουλειά που προσφέρει η Επιτροπή, η Αποστολή Επιτήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Και συμφωνώ με αυτά που είπε η Πρόεδρος που θέλησε να ενθαρρύνει τους συναδέλφους να επισκεφθούν τη Γεωργία και να ε, συμμετάσχουν στην αποστολή αυτή να επισκεφτούν επιτόπου συγκεκριμένες περιοχές. Τον Ιούνιο είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ το, τα διοικητικά σύνορα και να ε, δω επιτόπου το τι ακριβώς προσφέρει αυτή η επιστολή, αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα πει την ευκαιρία ε, με τα ίδια μου τα μάτια να δω ακριβώς ε, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τα διοικητικά σύνορα με την Απχαζία. Υπάρχουν χένουσες πληγές από τις εχθρότητες, αυτό μπορεί να το δει ο καθένας και μπορείς επίσης να δω και τα αποτελέσματα του τι είναι η συνεχιζόμενη ε, κατοχή ε, εκτάσεων στη Γεωργία. Πολλές φορές ε, ξεχνάμε πολύ εύκολα το τι συμβαίνει, αλλά το να βρίσκεται εκεί και να βλέπει κανείς ε, τους ε, Ρώσους πολιτοφύλακες ή τους Ρώσους στρατιώτες να είναι επιτόπου και να παρακολουθούν την περιοχή. Πιστεύαμε ότι αυτό έχει περάσει, είναι ανοίξει το παλιτόν, αλλά δεν είναι αλήθεια, εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω την ε, απαρασάλευτη θάση Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εδαφική αικαιρότητα της Γεωργίας. Πρέπει επίσης να σας πω ότι με απασχολεί πάρα πολύ η περίφημη διαδικασία συνοριοποίησης αυτό αφορά στο σύνολο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχει ε, ολέθριες επιπτώσεις ε, στον ντόπιο πληθυσμό και αναγκάζει πολλούς να εγκαταλείψουν τις αισθήσεις τους. Κάθε μέρα που περνάει υπονομεύονται οι προσπάθειες και η επιτροπή, η αποστολή επιτήρησης είναι εκείνη που δίνει κάποια δύναμη στους ανθρώπους των ε, όμορων, των άμεσα γειτονικών περιοχών. Μία ελπίδα ότι κάποιος, εν πάση περιπτώσει, κάπως εποπτεύει την κατάσταση ασφαλείας ε, στην περιοχή τους. Ε, πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, είμαι ακράδαντα πεπισμένος ότι έχει φτάσει πια στιγμή η Ρωσία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 12η Αυγούστου του 2008 για την πάψη πυρός και τις συμφωνίες επίσης του Μαΐου του 2008 που προβλέπει να αποσύρει το σύνολο των δυνάμεών της και να επιτρέψει στην αποστολή επιχείρησης πρόσβαση σε όλες τις κατεχόμενες περιοχές. Με άλλα λόγια, απλά ε, συμφωνώ και επαυξάνω με αυτά που ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Αν κανείς λάβει όλα αυτά υπόψη του, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξει το εξή. Συστήνουμε στις αρχές της Γεωργίας να έρθουν σε επαφή με τους κατοίκους ε, που ζουν στις ε, κατεχόμενες περιοχές, στην Νότιο Οσετία και στην Απχασία και αυτό μέσα από μια ε, πολιτική δέσμευση, όχι απαραίτητα αναγνώρισης. Για μας που είμαστε συνομοθέτες, εναπόκειται πλέον η πρωτοβουλία στο να καταργηθεί η θεώρηση. Ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να δώσουμε στη Γεωργία κάτι που της αξίζει, μία απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Αυτό θα διευκόλυνε τις επαφές ανάμεσα στους πολίτες και θα βοηθούσε και τους ε, Γεωργιανούς, ε, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κατεχόμενα. Επίσης, συμφωνώ με αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος του Συμβουλίου που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα να προσφέρει την ε, υποστήριξή της ε, για την εδαφική αικαιρότητα της Γεωργίας μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα. Έτσι λοιπόν ε, προσφέρω την αμέριστη υποστήριξή μου στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολύ καλή δουλειά της. Σας ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε σε πολύ δύσκολες συνθήκες και ευχόμαστε να ευοδοθούν οι προσπάθειες της αποστολής. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καρίμ ε, και εγώ ε, συμφωνώ με αυτό που είπατε για την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή είναι και η δική μου η προσωπική άποψη. Συμφωνώ με αυτά που λένε και όλοι οι άλλοι άμεσα εμπλεκόμενοι. Τώρα λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση. Αν θέλετε μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήσεις. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει κάποιος ε, περιορισμός χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω στις ε, παρεμβάσεις σας να τηρείτε αυτό το χρόνο, να προσπαθείτε να είστε σύντομοι. Πρώτα απ' όλα ο κ. Μάκλη Γκάλα, ο συντονιστής του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τους κυρίους ε, ε, Ντίν, την πρέσβη την κυρία Ζαμπανάτσε, τον κύριο Γιανκάουσκα και τον συνάδελφο Κάλιμ. Νομίζω ότι εδώ όσον αφορά τα μεγάλα κυρίως κόμματα επικρατεί συμφωνία. Όλοι συμφωνούμε στην αξιολόγηση της κατάστασης, συμφωνούμε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάρχει επιτόπου εδώ και πολλά χρόνια. Κατά τη δική μου άποψη, ως έχουν τα πράγματα δεν μπορεί κανείς να περιμένει η ρωσική πλευρά να επιδείξει μια πιο φιλική προσέγγιση ως έχουν τα πράγματα σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την παρουσία μας επιτόπου και με τον τρόπο αυτό ε, να επιτύχουμε και διαφάνεια όπου είναι αυτό δυνατό να ζητήσουμε από τη Ρωσία να εφαρμόσει αυτά τα οποία έχει υπογράψει. Ο κύριος Γιανκάουσκας είπε ότι τα πράγματα προχωρούν, η κατάσταση εξελίσθησε. Και αν ήθελα να επιδείξω λίγο σαρκαστικό, ηρωνικό πνεύμα, ε, θα έλεγα ναι, πράγματι μετακινούνται οι πινακίδες προς τα μπρος. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ. Μπορεί κανείς ε, άραγε να αναφέρει έναν αριθμό τετραγωνικών χιλιόμετρων. Δηλαδή πόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα διεύρυνε η Ρωσία τα κατεχόμενα και πόσους ανθρώπους αφορά αυτό. Αναφέρθηκε ότι ε, πρέπει να διατηρηθεί η επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκονται στα κατεχόμενα. Μα πώς το φαντάζεστε αυτό. Δηλαδή ε, σε αυτά τα σημεία διόδου Πόσοι άνθρωποι κατ' ουσίαν μετακινούνται κάθε μέρα από τη μία και την άλλη πλευρά των συνόρων ή μήπως ε, εξαρτάται από την ε, απόφαση που λαμβάνεται επί καθημερινά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και αυτοί που έρχονται προς τη γεωργία μπορεί η γεωργιανή κυβέρνηση να τους ερωτήσει από πού παίρνει η κυβέρνηση οργία τις πληροφορίες της. Και βεβαίως ε, απομένει και το θέμα το πολιτικό. Δηλαδή αυτή η απαράδεκτη κατάσταση μήπως ε, θα έπρεπε να μας οδηγήσει εμάς να επιβάλλουμε κυρώσεις ε, έναντι των ανθρώπων που βρίσκονται στην άλλη πλευρά και οι οποίοι εργάζονται παράτυπα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ερώτημα πολιτικής φύσεως Δηλαδή, εγώ κατ' ουσίαν προτείνω να επιβάλλονται συγκεκριμένες κυρώσεις σε ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου. Ο κύριος Φρόιντ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και την ε, πρέσβυρα καθώς επίσης και τους δύο κυρίους ε, για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που ακούσαμε από όλους. Είναι πάντα εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο να λαμβάνουμε πληροφορίες για τέτοιου είδους σειράξεις οι οποίες έχουν παγώσει για χρόνια. Συνήθως ακούμε ε, νέα όταν ε, γίνεται κάποια έκρηξη ε, και στην Παλαιστίνη το είδαμε. Μας το είπανε, δεν μας δεν ασχολείστε μαζί μας όταν τα πράγματα είναι σχετικό ήρεμα. Ε, όταν ε, υπάρχει κάποια έκρηξη τότε και οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης όλοι στρέφονται προς ε, το σημείο στο οποίο έχει γίνει η κρίση. Αλλά φυσικά δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους κρίσεις έτσι ώστε να διαφερθούμε για τη γεωργία. Θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση Άκουσα τον κύριο Γιανκάουσκας και την κυρία Σαμπανάτσε και ανείχνευσα μία σχετικώς διαφορετική άποψη σχετικά με το, την ε, πορεία των πραγμάτων επιτόπου. Ε, αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι εσείς μας είπατε ότι κάθε μέρα γεωργοί, ε, παιδιά του σχολείου περνούν τα σύνορα και ε, από ό,τι καταλάβαμε αυτό που είπατε, δεν ελέγχονται ε, στο, σημείο που ε, περνούν τα σύνορα. Ενώ η κυρία Σαβανάτζα μας είπε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι επικίνδυνο να πάει κανείς από το ένα σημείο στο άλλο και να διασχίσει τα σύνορα. Ε, ρωτώ λοιπόν από το ένα χωριό στο άλλο μπορεί να πάει κανείς εύκολα, ε, υπάρχουν μικροί δρόμοι ε, ή πρέπει να περάσει κανείς από τα αυστηρά ελεγχόμενα σημεία διέλευσης των συνόρων. Αυτό ήθελα να καταλάβω. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ πολύ ο κύριος ε, Παρσομαρακιούρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλεσμένους μας και να τους και να συγχαρώ τους εκπροσώπους της Επιτροπής Επιτήρησης για την επιτυχία της Επιτροπής. Εγώ η σώμαση ε, διεπίστωσα την ε, εργασία σας και έχετε δίκιο όταν λέτε ότι είσαστε τα μάτια και τα αυτιά μας, τα μάτια και τα αυτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γεωργία. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται ένθεν και ένθεν της διοικητικής συνοριακής γραμμής. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και την πρέσβη της ε, Γεωργίας. Ε, μία ερώτηση. Ακούσαμε τι συνέβη μετά από τον... Ξέρουμε τι συνέβη μετά από τον πόλεμο. Έγιναν εθνωτικές ανταλλαγές και αδιάφορες αλλαγές οι οποίες έχουν ακόμα συνεχίζονται όπως συνεχίστηκε η κατοχή κάποιων περιοχών. Ε, όμως ε, καταλαβαίνω ότι ξεκινούν κάποιες ε, σχέσεις και με την Απχαζία όσον αφορά κάποιες επενδύσεις κυρίως. Κυρία Πρέσβη, ποια είναι η κατάσταση της κοινή γνώμης στην Απχαζία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν, η κοινή γνώμη, οι επιχειρηματίες θέλουν να επανενωθεί με την Απχαζία. Πώς είναι η κατάσταση. Και έχω και μία ερώτηση ε, για τον κύριο Γιάνν Κάουσκας. Αναφέρατε κύριε Γιάνν Κάουσκας ότι στην Απχαζία θα γίνουν ε, κάποιοι, κάποιοι έλεγχοι των ξένων. Ε, θέλετε να μας πείτε τι εννοείτε ακριβώς και τι σημαίνει στην πράξη και ποιος θα καλύπτεται από αυτή τη νέα νομοθεσία. Σε ευχαριστώ πολύ, Κριστιαν Έλλερ. Thank um, Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πω στην ε, κυρία Πρέσβη ότι ε, θα θέλαμε να κάνουμε την αποστολή στην ε, ε Τυφλίδα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε στα προγράμματά μας. Σε σχέση τώρα με αυτά που είπε και ο κύριος Κάουσκας ε, στην φάση υλοποίησης ε, ε, της Επιτροπής Επιτήρησης βλέπουμε ότι υπάρχουν διεθνείς διαγωνισμοί σχετικά με διάφορα θέματα όσον αφορά τα καύσιμα κυρίως αλλά ε, καταλαβαίνουμε ότι οι κανόνες ε, της, ε, της διαδικασίας του διαγωνισμού έχουν δημοσιευθεί, αλλά εδώ και ένα χρόνο δεν έχει προχωρήσει καθόλου η κατάσταση. Η Επιτροπή μας εδώ και το Κοινοβούλιο γενικά και στη φάση των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό ανέλαβε τη θέση ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει μια διευκόλυνση των κανόνων ε, των διαγωνισμών όσον αφορά τις ε, μη στρατιωτικές επενδύσεις γιατί η παρουσία στα σύνορα είναι ε, ένα, πολιτικό, σημαντικό σκέλος αυτής της Επιτροπής ε, Επιτήρησης ε, και επομένως ποια είναι η άποψή σας όσον αφορά αυτήν την ελαστικοποίηση κατά κάποιο τρόπο των κανόνων των διαγωνισμών και των προμηθειών. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Γιάρομης Μετίνα. E, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στους προσκεκλημένους. Όποιος θέλει να απαντήσει. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε τρεις βασικούς αγωγούς. Μπακού Τυφλίδας, αγωγός φυσικού αερίου, τον πετρελαγωγό και το τελευταίο τον τεράστιο ε, αγωγό από την Τυφλίδα φτάνει μέχρι την Τουρκία και έχω το εξής ερώτημα. πετρελαγωγός που τροφοδοτεί με πετρέλαιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες η αποστολή μεριμνά για την ασφάλεια αυτών των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μεταξύ άλλων, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη είναι η εξή. Πολλές φορές έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ δύσκολο να επιτηρηθεί η κατάσταση στην Νότια Οσετία. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες διαπραγμάτευσης με την διοίκηση είτε στην πλευρά της Νότιας Οσετίας είτε στη ρωσική πλευρά για να υπάρξει μια μόνη παρουσία στην Νότια Οσετία. Και αν αυτό έχει, ε, δεν έχει γίνει δεκτό, ποια ήταν ε, η αιτιολόγηση της άρνησης. Thank you. Ευχαριστώ. Μόντι. Oh, okay, <laughs> I'm sorry. I was just explaining that I'm um, due Έλεγα ε, ότι πρέπει να φύγω για να μιλήσω σε μια άλλη επιτροπή. Τέλος πάντων, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να προσθέσω ή μάλλον να επαναλάβω και εγώ, ε, όπως οι προλαλήσαντες, ε, τα συγχαρητήρια για το έργο που έχει επιτελεστεί αυτό που υπόθηκε επίση για την απελευθέρωση των θεωρήσεων με βρίσκει σύμφωνη. Τέλο, θέλω να κάνω ένα ερώτημα. Έχετε κάποια αιτήματα ενδεχομένω από πλευρά αποστολή σε εμά του ε, βουλευτέ. Η πρέσβη ε, είπε μέσω των διαχωριστικών αυτών γραμμών ABL μίλησε για ενίσχυση των επαφών ενίσχυση των διασυνδέσεων των κοινοτήτων που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά αυτών των γράμμων. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ και με αυτή την παρέμβαση. Ολοκληρώνει το κατάλογο των ομιλητών και θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους μας με τη σειρά που έλαβαν πρώτο το λόγο ε, και πριν το λόγο να απαντήσουν. Κύριος Ντίν λοιπόν καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου για τις ε, δημόσιες προμήθειες και τις προκλήσεις ή διαγωνισμοί. Σίγουρα είναι πρόκληση για την αποστολή επιτήρησης το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε και πάντως, πάντα εκεί ακροβατούμε. Είναι λίγο διαφορετική αυτή η αποστολή επιτήρησης. Πρώτο ανεπτύχθη την 1η Οκτωβρίου. Είχαν συμφωνηθεί μόλις 28, 22 μέρες πριν ε, κάποια εκτελεστικά μέτρα. Και ήταν πάρα πολύ σύντομο το διάστημα και έπρεπε να παράσχουμε οχήματα, προσωπικό, ε, κομπιούτερ κτλ. κτλ. Βέβαια έχουν εξελιχθεί τα πράγματα από τότε, από το 8 δηλαδή. Έχουμε και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση από την Κομισιόν όχι ότι παρακάμπτουμε πράγματα, απλά είμαστε πιο εστιασμένοι πλέον και για τα οχήματα και για μεγάλα εξαρτήματα. Έχουμε και άλλες συμβάσεις επίσης. Έρχομαστε έτσι σε επαφή με κάποιους προμηθευτές. Αλλά πάντοτε επιδεικνύουμε τη δέουσα οικονομική σύνεση και διεκπεραιώνουμε γρήγορα, αλλά σεβόμενοι τους κανόνες. Ε, τους διαγωνισμούς. Ε, σε ό,τι αφορά την αποθήκη, το warehouse ε, που θα σας παρουσιάσουμε, ελπίζουμε οι δυνατότητες και η εντολή του να αναπτυχθεί στο μέλλον για να μπορούμε εκεί να αποθηκεύουμε αλλά και να κάνουμε και εργασίες βελτίωσης και εξυγχρονισμού του εξοπλισμού μας, οχημάτων και άλλων και άλλο εξοπλισμό. Επίσης πρόσβαση στα θωρακισμένα οχήματα είναι σημαντικό για την αποστολή. Έχουμε αρκετά οχήματα, έχουμε τα διάφορα θέατρα επιχειρήσεων. Θα φέρουμε οχήματα και από το Αφγανιστάν, ίσως το 2016 ελπίζουμε να έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία για να έχει τον ακατάλληλο εξοπλισμό η Γεωργία. Προσπαθούμε δηλαδή και νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να μετριάσουμε τους περιορισμούς. Έχουμε εξελίξει τον τομέα λοιπόν των διαγωνισμών, ε, της αποθήκης, της ε, σύναψης ε, συμβάσεων. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον εξοπλισμό μας και νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει από το 8 και μετά. Ευχαριστώ λοιπόν ο κύριος Γιάν Κάουσκας. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω ένα ερώτημα που είχε να κάνει με τον αντίκτυπο των συμβάντων στα δύο χωριά ε, το καλοκαίρι πέρυσι και αν μπορούμε να υπολογίσουμε τον αντίκτυπο αυτό. Εμείς εξετάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά την κατάσταση και το ότι συνέβη. Από τα δύο χωριά μιλάμε για 153 ανθρώπους, αγρότες, μέχρι πέρυσι μπορούσαν να καλλιεργούν την περιοχή των 58 εκταρίων μέχρι πέρυσι το καλοκαίρι. Πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο τη Φλίδας Γκόρη. Και βλέπετε, αν ε, οδηγείτε σε αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, τη βλέπετε αυτή την περιοχή. Τι έγινε όμως, μεταφέρθηκε η πινακίδα κατά 1,2 ε, χιλιόμετρα νοτίως προς τον αυτοκινητόδρομο. Δεν ήταν εκεί πριν. Αν άλλαξαν οι γραμμές, όχι δεν άλλαξαν. Όμως η συγκεκριμένη περιοχή καλλιεργείτο από άτομα τα οποία ζούσαν σε ένα, ε, στην επικράτεια που πάντοτε διαχειριζόταν από την δική του, από την τυφλίδα. Και η άλλη πλευρά αναφέρεται ε, στη γραμμή, στο χάρτη του 1984 και όμως δεν υπάρχει σήμανση. Τι έγινε λοιπόν. Μεταφέρθηκε, μετακινήθηκε η πινακίδα και είπαν σε αυτού του ανθρώπου ότι δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη γη σα, που είχαν και όμω τι καλλιεργίε του. Με την ενεργοποίηση του hotline ε, και ξεκινήσαμε και τι ε, συζητήσει μα, τι συνομιλίε μα στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού πρόληψη συμβάντων, καταφέραμε λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί πλέον να μπορούν έστω τη συγκομιδή τους να την ανακτήσουν, αλλά από την 1η Νοεμβρίου της περσίνης χρονής δεν έχουν πλέον πρόσβαση σε αυτήν την περιοχή. Αυτοί που είχαν λοιπόν τη γη και ήταν ε, για την επιβίωσή τους κρίσιμο αυτό, ε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν συνέπειες σίγουρα. Τώρα, τι γίνεται με τους σταθμούς διέλευσης. Μάλλον δεν τα είπα καλά. Ναι, φυσικά και υπάρχει δυνατότητα διέλευση. Στο θέατρο της Νότιας Οσετίας ε, έχουμε καταγράψει πάνω από 400 διελεύσεις την ημέρα. Στην Απχαζία ο αριθμός είναι μεγαλύτερος ακόμη. Κάθε μέρα βλέπουμε δύο με τρεις χιλιάδες ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται. Στην Νότια Σετία έχουμε ένα σημαντικό σταθμό διέλευσης και μόνο αυτοί που επέλεξαν να ζήσουν ε, στην κοιλάδα Χαμπόρη, στην Νότια Σετία, αυτοί έχουν ειδικέ άδειε. Όποιοι ε, επέλεξαν να ζουν εκεί και αυτοί μπορούν να περάσουν στη διοικητική επικράτεια της Τυφλίδας. Μία, ε, ε, ένα χρόνο ισχύει αυτή η άδεια. Έχουν κάποιοι λήξει το 14-15 θα λήξουν φέτος, αλλά έχουν ε, υπόψη τους οι άνθρωποι αυτοί το τι ισχύει και επαναλαμβάνω δεν πήραν όλοι ετούντες. Μόνο όσοι έχουν επιλέξει να ζουν εκεί. Τώρα Υπάρχουν κάποιες τοπικές διευθετήσεις για τους κατοίκους κάποιων χωριών. Αλλά η πρόσβαση για όλους τους άλλους ότι είναι πολύ περιορισμένη. Τώρα στην Απχαζία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πρέπει κάποιος να έχει ειδικά έγγραφα στη διάθεσή του για να μπορεί να περάσει. Και μόνο όσοι ζουν ε, στην περιοχή του Γκάλι. Και όχι όλοι. Δεν έχουν όλοι έγκυρα έγγραφα. Γιατί κάποια ε, μπορεί να σαν κάποια ζημιά. Κάποιοι μπορούν να περάσουν από κάποιες ανεξέλεγκτες, ε, ε, από μη ελεγχόμενες περιοχές μέσω του ποταμού Γκόρη για παράδειγμα και μάλιστα έχουμε και πνιγμούς. Από μη ελεγχόμενες περιοχές προσπαθούν να περάσουν ε, ορισμένοι, αλλά μπορεί να τους συλλάβουν οι αρχές που επιτηρούν και να τους επιβληθεί πρόστιμο. Για τα σχολεία. Όταν τα παιδιά ε, δεν τους επιτρέπεται να περάσουν στα σχολεία. Έχουμε πολλές φορές ε, τέτοια επεισόδια με, το, με τη μέθοδο της hotline αυτής της γραμμής μπορού. Προσπαθούμε να επιλύσουμε την κατάσταση και δυστυχώς τα πράγματα δυσκεραίνονται κάθε, σχολικό, κάθε σχολική χρονιά όλο και περισσότερο. Είναι όλο και πιο δύσκολο επίσης ε, να περάσει κάποιος για να επισκεφθεί το νεκροταφείο στο οποίο θα μένει συγγενής του. Που ήθεστε να γίνονται τέτοιες επισκέψεις το Πάσχα για παράδειγμα. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, ε, μάλλον ετησίως. Για παράδειγμα, στην διαχωριστική ε, συνορική γραμμή της Νότιας Οσετίας. υπάρχει ε, μια ε, γραμμή που έχει περιφραχθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πέρασει ο κόσμος. Είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Για τον νόμο περί αλλοδαπών. Έχουμε το σχέδιο στη διάθεσή μας και το μελετούμε. Θα ισχύσει από 1η Απριλίου και μετά αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά ήδη διαβάζοντάς το βλέπουμε ότι όσοι δεν είναι υπήκοοι της Αμπχαζίας δεν θα έχουν δικαίωμα δυνάμει αυτού του νόμου. να συμμετέχουν, να ψηφίζουν ούτε στις τοπικές ούτε στις εθνικές εκλογές. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ιδιοκτησία. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το νόμο και παραμένει ανοιχτό αυτό το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους διαγωνισμούς, νομίζω απάντησε ο διευθυντής και Ντίν. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις διαδικασίες. Μέχρι στιγμής δεν επηρεάστηκαν οι δικές μας επιχειρήσεις. Αν παρακολουθούμε τους αγωγούς, αν τους επιτηρούμε, ξέρουμε από πού περνά ο οδηγός Μπακού Σούψα. Εκεί μπήκε μια πινακίδα πέρσι το καλοκαίρι. Η British Petroleum είναι η διαχειρίστρια εταιρεία. Η εταιρεία αυτή παρακολουθεί λοιπόν. Σε κάποια σημεία χρειάζεται λιγότερη, σε άλλα περισσότερη επιτήρηση. Μπορείτε εσείς ίσως να απευθυνθείτε στην ΠΠ γιατί αυτοί επιτηρούν αυτό τον αγωγό. Σε ό,τι αφορά τώρα τι κάνουμε με τους Ρώσους και τους ε, Οσετούς. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε ένα διάλογο σε τοπικό επίπεδο με τους τοπικούς ε, φορείς ασφάλειας. Έχουμε και το IPRM κάθε μήνα, έχουμε και τη Γενέβη. Έχουμε λοιπόν συνεχή διάλογο και αυτό βοηθάει. Βοηθάει να επιλύονται κάποια από τα προβλήματα και να έχουμε κάποια πρόοδο. Βέβαια είναι περιορισμένη όπως είπατε σωστά. Ευχαριστώ και εδώ σταματώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιανκάσκας. Η κυρία Πρέσβης παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου υποβάλλατε. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σημεία διέλευσης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι συμφωνούμε, δηλαδή κατά τη δική μας άποψη η κατάσταση είναι η εξή. ότι τα σημεία διέλευσης, ε, εκεί τα πράγματα είναι πολύ περίπλοκα, γιατί πολλές φορές εφαρμόζονται ταπεινωτικές ε, ε, πρακτικές και μπορεί να συμβεί και κάποιο δυσάριστο γεγονές. Είπατε ότι πολλές φορές συμβαίνει κάτι απρόπτω αλλά ε, δεν ξέρει κανείς κάθε μέρα τι θα συμβεί. Μπορεί κάποιος να συλληφθεί χωρίς λόγο. Ε, αυτά τα τυχαία γεγονότα σε μια ευαίσθητη κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνα. Υπάρχουν απαγωγές, ε, υπάρχουν παράνομες κρατήσεις. Ε, αυτά προφανώς και επηρεάζουν και την κατάσταση στην τύφλιδα και δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Σε μια ιδανική περίπτωση, εάν υπήρχε μεγαλύτερη ευελιξία στα σημεία διέλευση. Ε, θα είχαμε μια ε, τελείως διαφορετική σύγκρουση. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν ε, αυτά τα φράγματα, αλλά αν υπήρχε πιο ελεύθερη διέλευση, αυτό θα επηρεούσε πάρα πολύ τη φύση της σύγκρουσης. Και νομίζω ότι σκόπιμα υπάρχουν αυτά τα σειρματοπλέγματα. Τώρα, όσον αφορά ε, την διάθεση που επικρατεί και κυρίως όσον αφορά το θέμα της Απχαζίας, ποια είναι γενικότερα, ποια είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ε, η δική μας ε, η πολιτική έχει ως στόχο στη συμμετοχή, στη δέσμευση. Και στόχος μας επίσης είναι να ε, έχουμε ε, στην Απχαζία ενδιαφερόμενους πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται να έχουν κάποια ένωση με τη Γεωργία. Και να επανέλθει ένα διεθνές νομικό πλαίσιο. Αυτό να αναγνωριστεί και να αναγνωρίζονται οι άνθρωποι ως πολίτες ενός εύρυθμα λειτουργούντος κράτους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το επιτύχουμε αυτό, υπάρχουν διάφορες δύο επικοινωνία. προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί μπορούμε για να τους δείξουμε πώς εξελίσσεται η γεωργία. Δηλαδή, ε, πώς ε, οι προτεραιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, μετατρέψει τη χώρα και πώς η αλλαγή αυτή έχει γίνει ελκυστική ε, και για τους ε, πολίτες. Ε, έτσι λοιπόν η κατάργηση απελευθέρωση των θεωρήσεων αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Θα είναι ένα μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αναγνωρίζει την πρόοδο της Γεωργίας και επίσης ένα πολύ σημαντικό ελκυστικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για οικοδόμηση εμπιστοσύνη και για να προσελκυστούν οι πολίτες και από την άλλη πλευρά. Όσον αφορά στις ε, συμφωνίες ε, ενσωμάτωσης ή ε, σύνδεσης, όταν αυτές συζητήθηκαν, υπήρξαν διαφορετικές αντιδράσεις στην Απχαζία. Οι πολίτες ήταν διχασμένοι, ήταν, υπήρξαν αρκετά αρνητικές και αρνητικές αντιδράσεις για πάρα πολλούς. Αυτό ήταν πολύ προχωρημένο και υπήρχε ο ουσιαστικός κίνδυνος η σύνδεση, οταν αυτες συζητηθηκαν υπηρξαν διαφορετικες αντιδρασεις στην απχαζια οι πολιτες ηταν διχασμενοι ηταν υπηρξαν αρκετα αρνητικες και αρνητικες αντιδρασεις για παρα πολλους αυτο ηταν πολυ προχωρημενο και υπηρχε ο ουσιαστικος κινδυνος η απχαζια de να ενσωματωθεί ε, στην Ρωσική Ομοσπονδία, κάτι το οποίο όμως δεν επιθυμούσαν. Πάντως υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες και οι ακόλουθες, οι διάδοχες ε, συμφωνίες είναι εκείνες ε, οι οποίες συζητούνται και θα υπογραφούν. Ανησυχούμε λοιπόν ότι πράγματι αυτή είναι μια διαδικασία σταδιακής προσάρτησης, θα γίνουν όλα πολύ ήπια, πολύ σιωπηρά. Είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσει κανείς με αυτόν τον τρόπο την ε, προσοχή και το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας, αλλά ε, μας ανησυχεί γιατί φοβούμαστε ότι αυτό θα παρουσιαστεί ως ένα τετελεσμένο γεγονός. Όσον αφορά τώρα την εθνοκάθαρση, η εθνοκάθαρση πράγματι έχει υπάρξει κυρίως όσον αφορά τους Γεωργιανούς και χωριά στη Γεωργία τα οποία καταστράφηκαν σκόπιμα, ε, κάηκαν. Ε, δεν έχουμε καμία πρόοδο ε, σχετικά όσον αφορά στην επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων και είναι πρόβλημα. Δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο το να επιτευχθεί η πρόοδος. Όσο λοιπόν δεν επιστρέφουν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι, μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι παραμένει γεγονός η εθνοκάθαρση. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που επικρατεί. Δυστυχώς η συνοριοποίηση που συζητήθηκε, η συνοριοποίηση αυτή δεν βοηθάει την κατάσταση και δημιουργεί τον κίνδυνο να εμφανιστούν και άλλοι εσωτερικά εκτοπισμένοι γιατί όπως αναφέρθηκε ε, υπάρχει ο φόβος να μην έχουν πρόσβαση στη γη την οποία καλλιεργούσαν. Υπάρχουν περιπτώσεις που. Μία γυναίκα, ε, με μία οικογένεια ξύπνησε ένα πρωί και ξαφνικά είδανε ε, στην αυλή του είχε γερθεί σειρματόπληγμα και δεν μπορούσαν να πάνε στο χωράφι του. Ορισμένε οικογένειε αναγκάστηκαν να φύγουν, να εγκαταλείψουν τι αιστείε του ε, και αυτό ως αποτέλεσμα των κινήσεων που σας ανέφερα. Στην Απχαζία αυτές οι συμφωνίες και περαιτέρω περιορισμοί ε, πρόσβασης σε θέματα επικότητας, άδεια παραμονής, ε, ό,τι δηλαδή είναι απαραίτητο για να ζει κανείς ε, ως άνθρωπος με αξιοπρέπεια, δηλαδή πρόσβαση σε ιδιοκτησία, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Υπάρχουν όλο και μεγαλύτεροι περιορισμοί στη Ρωσία και στην Απχαζία για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και αυτό δημιουργεί πίεση σε όσους παραμένουν στη γη τους και φοβούμεθα ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των εσωτερικών εκτοπισμένων. Όσον αφορά αυτήν την κατάσταση, δυσάρεστα τα νέα. Επίσης ε, και η πρόσβαση από το εξωτερικό, πολύ περιορισμένη. Ο, ε, είπατε, είπατε εκπροσώπηση, ο είπατος ε, επίτροπος ε, για τους ιστορικά εκτοπισμένους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι δύο θέλησαν να πάνε στην Απχασία, τους το αρνήθηκαν. Θέλουμε λοιπόν να υπάρξει μια διεθνής αξιολόγηση ε, της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα όσον αφορά τον Μπακού, ε, τον αγωγό Μπακού, τη φλίδα, τον ε, αγωγό πετρελαίου, 1600 μέτρα είναι αυτός ο αγωγός. Και αυτός τώρα επίσημα βρίσκεται στα κατεχόμενα. Την κατάσταση ελέγχει η BP. Όμως, για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται η στρατηγική σημασία αυτής της περιοχής και με τον τρόπο αυτό αυξάνεται γενικότερα η σημασία της περιοχής γιατί αυτοί οι αγωγοί έχουν σημασία όχι μόνο για τη Γεωργία αλλά όπως είπατε για τη σταθερότητα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam Ambassador. Now, Mr. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Καρύμ. Ένα-δυο σημεία ε, θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ε, τους ε, πανελίστες μας. Ο Μαρκ ρώτησε για ποιες περιοχές μιλάμε. Αν δεν σφάλω, μιλάμε για περίπου 63 χιλιόμετρα αγγυλωτού σύρματος, τέτοιου φράχτη δηλαδή σε συνεχή βάση και η ε, πρέσβης ε, με πολύ ε, αδρά χρώματα περιέγραψε τι συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις και θα ήθελα να πω και δύο λόγια σχετικά με αυτό που μας είπε ο κύριος Κεστούσης Γιανκάουσκας. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση ιατρικού προσωπικού ή για, για κάλυψη ιατρικών αναγκών. Σε πολλές περιπτώσεις η Επιτροπή Επιτήρησης ε, ε, βοηθάει την διέλευση ασθενοφόρων που διακομίζουν ασθενείς. Ε, κατά τα υπόλοιπα μπορώ να συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Πρέσβη. Ε, η Γεωργία νομίζω ότι έχει ήδη δείξει δείγματα γραφής ε, της προσήλωσης της στην Ευρώπη και της αναγνώρισης της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αναγνωρίζεται μέσω της νέας κατάστασης όσον αφορά του, τις θεωρήσεις της ταξιδιωτικές, τις βίζες δηλαδή και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για τη Γεωργία λειτουργεί αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της ευελισσίας διατάξεως με μία παρατήρηση. Εγώ συχνά έχω επισκεφθεί ε, εδώ και πολλά χρόνια την περιοχή. Το 2009, το 2010 ξεκίνησα να ε, επισκέπτομαι ε, τις τις ε, εγκαταστάσεις της IDP στην Γεωργία και πραγματικά τα πράγματα είναι πολύ καλά. Πρέπει να σας πω ότι αυτοί που ζουν ε, στις περιοχές θέλουν να γυρίσουν πίσω. Είναι προφανές. Είναι προφανές. Ε, οι ε, εσωτερικώς εκτοπιστέντες θέλουν να επιστρέψουν. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις δικές μου επισκέψεις στο κέντρο αυτών των εσωτερικά εκτοπισμένων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφήσει πίσω οικογένειες, ε, βεβαίως μπορούν να τους επισκεφθούν, αλλά ε, όταν κανείς μιλήσει μαζί τους διαπιστώνει αμέσως ότι θέλουν να γυρίσουν στην Νότια Οσετία, στην Απχαζία Θεωρούν ότι αυτή είναι η γη τους. Είναι παραπάνω από προφανές. Κυρία Πρέσβη, κύριε κύριοι Ντίν και Γιάν Κάουσκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση η αποστολή της Επιτροπής μας τον Μάιο θα επισκεφθεί την Τυφλίδα και επομένως θα έχουμε και μία επιτόπου ενημέρωση επιπλέον. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, μην φύγετε. Αρχίζουμε αμέσως με την εξέταση του επομένου θέματος σημερισίας διατάξεων. Ευχαριστώ. Ladies and gentlemen, please be seated. Uh, we Παρακαλώ καθίστε γιατί θα ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. Όσο περιμένουμε και τον τρίτο μας ε, ομιλητή, ας ξεκινήσουμε ήδη τη συζήτηση. Ε, συζήτηση η οποία θα αφορά την κατάσταση ασφαλείας στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα ε, ε, σας πω ότι η κυρία Μάρτα Τσίγκαν, Διευθύντρια Αρμόδια για τη Στρατηγική ε, για τις γενικές υποθέσεις, Γενική Διεύθυνση Home, ζητά συγγνώμη, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί έχει μια σημαντική video conference με την Τουρκία θα έχουμε πάντως την ευκαιρία να ε, υποδεχθούμε έναν εμπειρογνώμονα από τη Γενική Διεύθυνση Home ε, και επομένως θα συζητήσουμε το θέμα χωρίς κανέναν περιορισμό. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον καθηγητή Φλόριαν ε, Τράουνερ, του Φράι Universität των Βρυξελών, του Ελεύθερου Πανεπιστημίου των ε, Βρυξελών. Θα έχουμε επίσης τον κύριο Άντρου Ράσπας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος εδώ της Γενικής Διεύθυνσης ΝΙΑΡ, θα έρθει. Η κυρία Μάρθα Τσίγκαν, όπως σας είπα, αντικαταστάσει από τον κύριο Μόρτον Μπέναντεκ, ο οποίος είναι έμπειρογνώμονας στη Γενική Διεύθυνση HOME. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν ε, πρώτα απ' όλα με την ε, παρέμβαση του ε, καθηγητού κυρίου Τρόνερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες διαφάνειες. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, κυρία Πρόεδρε, Έχω διάφορες ε, παρουσιάσεις όσον αφορά την ε, ε, παρούσα κατάσταση της ασφάλειας των, στα Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως σε σχέση με την προσφυγική κρίση. Θα ξεκινήσω με τις πολιτικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων. Έχουν υπάρξει αρκετές σημαντικές εξελίξεις τους τελευταίους μήνες, να μην πω τις τελευταίες μέρες η Βοσνία Ερζεγοβίνη υπέβαλε αυτή τη βδομάδα έτοιμα για την ένταξη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κωσυφοπαίδιο τον προηγούμενο Οκτώβριο υπέγραψε τη Συμφωνία Ειρήνευσης. Το Μαυροβούνιο ε, και η Σερβία προχωρούν επίσης ε, τις διαδικασίες ένταξης. Έχουν, έχουν κλείσει ήδη δύο κεφάλαια στο, στο Μαυροβούνιο, έχουν ανοίξει άλλα και στη Σερβία έχουν κλείσει δύο κεφάλαια. Το ζήτημα προκύπτει πλέον με την Φύρο, υπάρχουν νέες εκλογές για τον μη μήνα ε, Απρίλιο έχουμε πολλές διαμαρτυρίες ε, κατά του, της κυβερνήσεως του Νικολά Γκρουεύσκη, αλλά παρόλα αυτά ε, και, υπάρχει και η σαφή απειλή για μποϊκοτάρισμα των εκλογών από την αντιπολίτευση σε περίπτωση που δεν υπάρξει απελευθέρωση και ελευθερία έκφραση των μέσων ενημέρωσης. όσον αφορά τις όσον αφορά τις αποστολές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα θυμάστε ότι τον ε, Ιούνιο του 2016 λίγη ε, η αποστολή Ulex στο Κωσυφοπαίδιο, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να σκεφτόμαστε εάν οι αρχές είναι, του Κωσυφοπαιδίου είναι έτοιμες να αναλάβουν την κατάσταση. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2016 οι δικαστές του, της αποστολής Ulex έχουν ε, αποδώσει κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου σε Σέρβους πολιτικούς. Το ερώτημα λοιπόν όπως έλεγα και προηγουμένως είναι εάν και κατά πόσον ε, οι αρχές ε, του Κωσυφοπεδίου είναι έτοιμε να αναλάβουν την κατάσταση. Η ιδέα ήταν τον προηγούμενο Δεκέμβρη να υπάρξει επιμήκυνση για ένα χρόνο. Συζητήθηκε το θέμα και στα Ηνωμένα Έθνη. Ο Βαλεντίνο Κόφσκο ε, ε, ανέφερε ότι ε, υπάρχει ανάγκη για εξακολούθηση αυτής της αποστολής. Η Republica Σέψκα ανέφερε ότι θα διενεργήσει δημοψήφισμα για τα θέματα αυτά και επομένως μέχρι τώρα οι πολιτικές ε, ε, σχέσεις ε, λαμβάνουν χώρα υπό τον, μέσα στις γεωπολιτικές δυναμικές και την ανάλυση και του ρόλου του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Το Μαυροβούνιο έλαβε πλέον επίσημη πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν μιλάμε για, το, για τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Ε, ο Πρωθυπουργό Μίλο Τσογκάνοβιτς κατηγόρησε την Ρωσία ότι υποδαβλίζει διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα κατά ε, της ένταξης αυτής. Ε, το Μόσταρ είναι κατά της, ε, ε, της ένταξης στο ΝΑΤΟ και θεωρεί ότι η διεύρυνση του ΝΑΤΟ σε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα αποτελέσει μεγάλη πρόκληση για την Ρωσία. Είναι γεγονός ότι τα Δυτικά Βαλκάνια ε, υπάρχουν πολλές ε, συμφωνίες ε, για την ενέργεια και δημιουργούνται προβλήματα όσον αφορά τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες, κυρίως σε σχέση με μέτρα τα οποία έχει αναλάβει ή και έχουν εφαρμόσει οι Ηνωμένε Πολιτείες, κυρίως μετά την κατάληψη της Κρυμαίας. Η Σερβία ε, εξεκολουθεί να ε, κρατάει ε, ουδέτερη στάση και εξακολουθεί να έχει και σχέσεις και με την Ρωσία. Τώρα, θέματα καθαρά ασφάλειας, το θέμα των αλλοδαπών, των ξένων μαχητών. Η ISIS ε, έχει ξεκινήσει συγκεκριμένες στοχευμένες δράσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, ε, κυρίως όσον αφορά ε, νέους μαχητές από την Βοσνία και το Κωσυφοπέδιο. Να μην λησμονούμε ότι υπάρχουν ήδη και ακόμα μάλλον και κάποιοι βετεράνοι από τους πολέμους της περιοχής Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, περίπου 600 ξένοι μαχητές από την περιοχή έχουν ε, ε, συμπαραταχθεί με τον ISIS ε, στην Συρία και περίπου 100 πιστεύετε ότι έχουν επιστρέψει στην περιοχή ποια είναι η πολιτική απάντηση στην πρόκληση αυτή. Ε, η κυβέρνηση της Βοσνίας έχει καταβάλει κάποιες προσπάθειες, αλλά ακόμα πολλές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ε, είναι καταγερματισμένη η προσπάθεια γιατί υπάρχουν 22 αστυνομικές υπηρεσίες με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες. Επίσης ε, δεν είναι σωστή η συλλογή δεδομένων όσον αφορά τους ε, ξένους μαχητές και τους ξένους μαχητές που έχουν επιστρέψει ε, γνωρίζουμε ότι η κατάσταση οικονομική είναι κακή και επομένως είναι εύκολο να υποθάλψει τέτοιου είδους ακραίες ε, καταστάσεις. Το Συμβούλιο Υπουργών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ε, έχει παρουσιάσει μία στρατηγική στο πρότυπο της στρατηγικής των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά το θέμα της των ξένων μαχητών έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό ε, των μαχητών. Ε, φτάνω τώρα στο τελευταίο τμήμα της παρουσίασής μου, δηλαδή ε, τα θέματα της ασφάλειας σε σχέση με την προσφυγική κρίση. 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν φτάσει στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση ε, το τελευταίο καιρό, εκ των οποίων 760.000 έχουν επιλέξει ε, την οδό των Δυτικών Βαλκανίων για να φτάσουν στην Ευρώπη. το μεγαλύτερο μέρος αυτών έχουν περάσει από τα επίσημα σημεία διέλευσης των ε, συνόρων. Σύμφωνα με τις ε, αρχές, με τα στοιχεία της ε, Frontex, τα 60% περίπου των προσφύγων που έφτασαν στα σύνορα της ΦΥΡΟΜ δεν είχαν ελεγχθεί. Από το Σεπτέμβριο του 2015 αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρχισαν ε, να ε, χτίζουν φράχτες ε, ή να ελέγχουν περισσότερο τα σύνορά τους και είναι πλέον σαφές ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη ελέγχου των εξωτερικών σύνορων. Αυτό κατέστησε σαφές και από τις εργασίες του Κοινοβουλίου αλλά και από τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα Δυτικά Βαλκάνια οπωσδήποτε είναι άμεσα ε, αναμεμειγμένα στην ε, ε, διαδικασία και Αυτό έχει συζητηθεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επικεφαλής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά τα, ε, υψηλή η αριθμή ε, των ε, προσφύγων που φτάνουν στα σύνορα. Ε, από τις διελεύσεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες, 99% ε, εξ αυτών ε, είχαν περάσει μέσω, της, μέσω του Αιγαίου. Η πρώτη εθνικότητα είναι η Σύρη και μετά Αυγανοί, Ιρακινοί κλπ. ποιοι είναι τώρα οι κίνδυνοι όσον αφορά την ασφάλεια και ποια είναι τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα ε, έχουν αρνητική επίπτωση στην ε, περιφερειακή σταθερότητα. Επομένως, το κύριο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να ε, αποφύγουμε την περιφερειακή ένταση σε περίπτωση που τα κράτη, τα βορειότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλείσουν τα σύνορά τους. Ε, άλλο ερώτημα είναι η ενδεχόμενη παρίσφρηση τζιχαντιστών ε, μέσα από την ροή ε, των προσφύγων. Ε, μετά από τις, ε, επιχειρη... μετά από τις ε, απόπειρες του Παρισιού του προηγούμενου Νοέμβρη κατέστησαν φές ότι ορισμένοι εκ των τρομοκρατών είχαν καταφέρει να παρισφρήσουν μέσα στις προσφυγικές ροές. Θα πρέπει να σταματήσει η ε, θα πρέπει να ελεγχθούν περισσότερο τα σύνορα, θα πρέπει ε, να ελεγχθεί περισσότερο η διαδικασία καταγραφής ε, των προσφύγων, κυρίως δε όσον αφορά κάποια σημεία πίεσης. Επίσης υπάρχει και το θέμα του τράφικινγκ είναι ένα θέμα ε, ε, για το οποίο ζητούν επιπλέον ε, πόρους η Frontex, η Europol και η Eurojust, αλλά και μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ αυτών. Υπάρχει επίσης και ένα νέο κέντρο για την για την ε, παράνομη εμπορία ανθρώπων που θα ανοίξει στα πλαίσια της Europol ε, τον Φεβρουάριο του 2016, αυτό το μήνα δηλαδή, ε, και ξέρουμε ότι τώρα πλέον η βάση δεδομένων για το θέμα της Europol περιέχει πάνω από 38.600 υπόπτους και μόνο για το 2015 είχαμε 10.000 επιπλέον ε, επιπλέον υπόπτους. Επίσης θα πρέπει ε, στο Αιγαίο να γίνει μια προσπάθεια να κλείσουν τα σημεία παράνομης ε, διέλευσης. Θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία με την Frontex. Βεβαίως αυτή τη στιγμή μετά από αίτημα της Ελλάδος έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο που θα συνεργαστούν στενά με την ε, Frontex, αλλά παρόλα αυτά ακόμα δεν είναι αρκετές ε, οι προσπάθειες ε, και εκπρόσωποι της Frontex αλλά και εκπρόσωποι της, για τους πρόσφυγες λένε ότι θα πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν χώρες επίσης όπως η Φύρομ ή όπως η Σλοβενία οι οποίες προτίθενται ή έχουν δηλώσει μάλλον την πρόθεση πρόθεσή τους να ε, ε, ε, ελέγξουν με αστυνομικά μέσα περισσότερο τα σύνορά τους. Αυτά ήταν τα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας υποβάλω και σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπεναντέκ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι εδώ. Ο διευθυντής μου δεν μπορούσε να έρθει, διότι όπως είπε η πρόεδρος, υπάρχει μια βιντεοδιάσκεψη με την Τουρκία. Εμείς από την Επιτροπή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την προσφυγική κρίση. Έπρεπε λοιπόν η διευθύντριά μου να ε, φύγει και είμαι εγώ να, εδώ. Να σας πω και εγώ τι κάνουμε στα Δυτικά Βαλκάνια, πώς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δράση μας από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσουμε τις πτυχέ ασφάλεια. Τέσσερα σημεία θέλω να αναφέρω. Πρώτον, είναι πολύ σημαντική ανταλλαγή πληροφοριών. Ενώ στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, ε, ποινικά στοιχεία, στοιχεία που έχουν να κάνουν την επιβολή του νόμου. Μεταξύ άλλων, οι τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού μας δίδαξαν ότι δεν τροφοδοτούσαν όλες οι χώρες το σύστημα πληροφοριών της Europol με πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους η αστυνομία, οι, οι υπηρεσίες ε, πληροφοριών για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να περνάνε από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις ε, λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος πληροφοριών είναι πρώτον να βελτιώσουμε τι λειτουργίε δυνατότητε και δεύτερον να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να τροφοδοτούν το σύστημα πληροφοριών τη Ευρωπόλ. Αυτό θα είναι ένα κόμβο ευρωπαϊκών στοιχείων και θα μπορούμε να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε ενδεχομένω τρομοκρατικέ δραστηριότητε εντό και εκτό Ένωση. Για τα σύνορα, τέσσερι από τι πέντε πλήν του κοσφοπεδίου, δηλαδή έχουν ε, επιχειρησιακές συμφωνίες με την Ευρωπόλ, Σερβία, δηλαδή Αλβανία, Φύρομ και Μαυροβούνιο. Και οι τέσσερις αυτές χώρες έχουν την τεχνική δυνατότητα λοιπόν τα ξενωμένες διαβαθμισμένες πληροφορίες να τις τροφοδοτούν στο σύστημα και να λαμβάνουν αντίστοιχε πληροφορίες από την Ευρωπόλ και αυτό είναι ελπιδοφόρα εξέλιξη για την ανταλλαγή τέτοιων πληροφοριών που είπε και ο Φλόρια. Παραδείγματο χάρη, σπαστικοποιημένοι μαχητέ που γυρίζουν από τη Συρία και πάνε στη Βοσνία, μπορεί να περνάνε στην Αλβανία. Σήμερα οι αλβανικές αρχέ μπορούν να διαβιβάσουν σε άλλε αρχέ επιβολή του νόμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτέ τι πληροφορίε. και αυτό που προσδοκούμε είναι ότι αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα βελτιώσει τον εντοπισμό τρομοκρατών που έρχονται από τη Συρία και το Ιράκ ή την ικανότητά τους ε, να μειώσουν ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, ε, να περιορίσουν τη δράση τους. Οι αρχές με αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Δεύτερο τμήμα. Ριζοσπαστικοποίηση, πώς μπορούμε να την προλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις προσπάθειές στον τομέα αυτό. Υπάρχει και ένα δίκτυο ευαισθητοποίησης κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Τον Οκτώβριο άνοιξε αυτό το δίκτυο με στόχο για την πρόταση της Επιτρόπου Μάλστρομ το 2011, ε, να έρθουν σε επαφή με τους επαγγελματίες. Εσείς που είστε χαράκτη πολιτικής ξέρετε τι θα πει ρίζοσπαστικοποίηση. Οι επαγγελματίες πρέπει να μάθουν. Δηλαδή οι σοφρονιστικοί φύλακες, ε, οι εκπαιδευτικοί, όσοι έρχονται σε επαφή με τοπική κοινωνία. Νομίζω 2.000 άνθρωποι από διάφορα κρατημέλη εντάσσονται σε αυτό το δίκτυο και ανταλλάσσουν πληροφορίες για το πώς μπορούν να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση και τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών σε, ε, στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, θα μπορούσε να ανοίξει αυτό το δίκτυο κατά περίπτωση και σε τρίτες χώρες, θα μπορούσαν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, κάποιες από αυτές, να είναι καλές υποψήφοι. Υπάρχει κέντρο αριστείας, στο οποίο μπορούν να επωφεληθούν και αυτές οι χώρες. Έχουμε την πρωτοβουλία καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Με ήπια μέτρα ξεκινήσαμε ανταλλαγή πληροφοριών, εκπαίδευση συμμετοχή των αρχών επιβολή νομοθεσία των χωρών αυτών σε κάποιε από τι ευρωπαϊκέ δραστηριότητε. Υπάρχουν όμω και κάποια πιο ε, αποφασιστικά μέτρα, ανταλλαγή πληροφοριών και επιχειρησιακή δράση ε, σε ιδεατή περίπτωση από τις αρχή επιβολή του νόμου, αυτό όμως σε μεταγενέστερο στάδιο. Αργότερα θα έχουμε μια διάσκεψη. Είχαμε και τον Οκτώβριο μια πολύ πτυχημένη διάσκεψη, ήρθαν πολλοί και το 2016 θα έχει συνέχεια αυτή η πρωτοβουλία. Τρίτο σκέλος. Το ανέφερε και ο Φλόρια στην παρουσίασή του. Η παράτυπη μετανάστευση πάντα από την πτυχή της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας κύκλος πολιτικής ε, κατά του οργανωμένου κλίματος. Έχουμε τη μόνη επιτροπή COSI για την εσωτερική ασφάλεια στο Συμβούλιο, μια επιτροπή που σχετίζεται με το PSE και την εσωτερική ασφάλεια. Και το βασικό πλαίσιο που διέπει όλες αυτές τις δραστηριότητες κατά ε, κάποιων ε, πρόσφορων εδαφών για την τρομοκρατία είναι δύο ομάδες δράσης, συμμετέχουν τα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο την, παράνομη, την ε, πρόληψη της ε, παράτυπης μετανάστευσης και επίσης η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, για την προσφυγική κρίση διαβάζεται κάθε μέρα στον τύπο. Τι όμως περιγράφω εδώ. Μιλάω για μια επιχειρησιακή ουσιαστικά δράση με στόχο εταιρείε ε, ε, μεταφορών, συγκοινωνιών, ε, πούλμαν, που μεταφέρουν ή διευκολύνουν τη μετακίνηση κάποιων εντός της περιοχής της, του Σέγγεν. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε ύποπτους ή χρήση πλαστών, εγγράφων. Τα χρησιμοποιούν συχνά εγκληματίε για να διευκολύνουν την είσοδο υπηκών τρίτων χωρών στην Ένωση, τους δίνουν μια ευρωπαϊκή ταυτότητα ή κάποια άδεια εισόδου που τους επιτρέπει να μπορούν να παραμείνουν για μακριό χρονικό διάστημα. Και είναι πλαστά αυτά τα έγγραφα. Τέτοιου είδους δραστηριότητες προσπαθούμε να εντοπίσουμε από πλευράς Ευρωπόλ με τη συμμετοχή και κρατών των Δυτικών Βαλκανίων. Να μην σας πω πόσο επιτυχημένη ήταν αυτή η προσπάθεια. Ε, σίγουρα δουλεύουμε οι αρχές επιβολής του νόμου. Ε, κάνουν ό,τι μπορούν. Μια άλλη μας ενέργεια, μια άλλη δράση αφορά κυρίως τις ε, εγκληματικές συμμορίες που έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια για να διαπράξουν εγκλήματα κατά της περιουσίας, κλοπές, ληστείες, κλοπές ε, οχημάτων. Πάντα διοσυνοριακά γίνεται αυτό. Πολλά κράτη-μέλη αντιλήφθηκαν ότι είναι σημαντικό και οι ομόλογοι της Δυτικά Βαλκάνια να συνεργαστούν. Είμαστε σε πρώιμο στάδιο υλοποίηση και σε αυτή την περίπτωση, αλλά είναι ένα project στο οποίο συμμετέχουν τα Δυτικά Βαλκάνια. Τέλος, πυροβόλα όπλα. Το ανέφερε ο Φλόριαν. Διδαχθήκαμε πολλά μετά τις δημοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού. Όπως ότι ορισμένες από τις εκρηκτικές ύλες που χρησιμοποίησαν στο Παρίσι τρομοκράτες ήταν αυτοσχέδιες. Οι πρόδρομες ουσίες δε σε πολλές περιπτώσεις είχαν έρθει, ε, ήταν αποτέλεσμα λαθρεμπορίου και είχαν έρθει από τα Δυτικά Βαλκάνια, στα οποία υπάρχει και ένα μεγάλο οπλοστάσιο μετά από τον πόλεμο της δεκαετίας του 1990 και πολλά από αυτά τα όπλα πέφτουν στα χέρια εγκληματιών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προσπαθούμε να κάνουμε στον τομέα αυτό ήπια μέτρα προς το παρόν έχουμε. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης στο οποίο συμμετέχουν Ευρωπαίοι επαγγελματίε και ε, οι ομόλογοι τους από τα Δυτικά Βαλκάνια. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε, να αποσυναρμολογήσουμε όπλα, αλλά και να ε, εντοπίσουμε τις αποθήκες, τα απλοστάσια αυτά, που υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι πολύ, πολλά υποσχόμενος και αυτός ο τομέας. Δύσκολα μπορεί κανείς να κανείς να πει βέβαια ακόμη γιατί είναι επιχειρηματικέ οι πληροφορίε. Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε το μέγεθο επιτυχία, αλλά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, οι κυβερνήσει από τα Δυτικά Βαλκάνια στο μεγαλύτερο βαθμό συμμετέχουν και είναι και προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τις τρομοκρατικέ επιθέσεις του Παρισιού. Θέλουμε να περιορίσουμε την εμπορία όπλων από τρίτες χώρες. Είναι προτεραιότητα. Για την προσφυγική κρίση. Καλό θα ήταν ίσως να ακούσω τα δικά σας ερωτήματα γιατί η δική μας προοπτική είναι λίγο διαφορετική ε, σε σχέση με τις, προοπτικές, ε, με προκλήσεις ασφαλείας. Η διαχείριση των συνόρων σίγουρα είναι ένας τομέας, μπορούμε να τον συζητήσουμε σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά θα ήθελα πρώτα να ακούσω τις δικές σας ερωτήσεις και να απαντήσω μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος Ράσουμπας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, ζητώ συγγνώμη από εσάς και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής γιατί καθυστέρησα να έρθω. Ε, δεν μπόρεσα να ακούσω τους ε, προλαλήσαντες. Ελπίζω λοιπόν να μην επαναλάβω αυτά τα οποία έχετε ήδη ακούσει. Και γι' αυτό, ε, για να περιορίσω και τι δυνατότητε να επαναλάβουμε, ε, θα είμαι σύντομο. Δεν είμαι εμπειρογνώμονο σε θέματα ασφάλεια, αλλά μου ζήτησαν να έρθω εδώ για δύο λόγου. Κυρίω για να δώσω μια πιο ε, σφαιρική άποψη τη πολιτική τη Γενική Διεύθυνση, κυρίω για τα Δυτικά Βαλκάνια. Και δεύτερον, για να δείξω αυτά που μόλι ελέγξαν, δηλαδή το θέμα των μεταναστευτικών ροών από τα Βαλκάνια. Αυτό είναι κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα του τελευταίου οκτώ μήνε ε, και νομίζω θα μας απασχολήσει για αρκετό καιρό ακόμα. Όσον αφορά λοιπόν μια επισκόπηση της ε, ε, θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κομισιόν για τα Δυτικά Βαλκάνια. Κοιτάξτε, πρόκυψε, υπήρξε μια ουσιαστική αλλαγή πριν από 3-4 χρόνια όταν δηλαδή αντί για την τεχνοκρατική άποψη που είχαμε ε, σε παλαιότερες διευρύνσεις δηλαδή τι γίνεται με το κοινοτικό κεκτημένο και τι κάνει η χώρα γι' αυτό τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε ε, και δίνει σημασία στα βασικά ε, τα βασικά τι σημαίνει είναι θέματα διακυβέρνησης μάχης κατά της διαφθοράς θέματα που αφορούν στο κράτος, ε, μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Ίσως όλα αυτά να φαίνονται περίπλοκα, αλλά μας ενδιαφέρει και η διαχείριση των ε, δημόσιων οικονομικών. Διότι θεωρούμε ότι αν κάποιος επιθυμεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο έγκλημα στα Βαλκάνια και όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στους πολιτικούς και το οργανωμένο έγκλημα στα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτό δεν εκπλήσει κανένα. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο είναι παρακολουθώντας τη ροή του χρήματος, εξετάζοντας πιο ουσιαστικά τη νομιμοποίηση από έσοδα ε, εγκληματικών πράξεων, το ξέπλυμα του χρήματος όπως λέμε. Η αντίδραση λοιπόν γενικότερα του κόσμου ήταν ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για θέματα οργανωμένου εγκλήματος και ασφάλεια στα Βαλκάνια, διότι αυτά δεν επηρεάζουν μόνο τις ίδιες τις χώρες, αλλά και γενικότερα τη διεθνή κοινότητα. Και γι' αυτό λοιπόν οι ε, συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων παρακολουθούν εκ του σύνεγγυ το τι διαδραματίζεται. Ένα λοιπόν από τα θέματα που ενδιαφέρουν είναι το ότι υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στα Βαλκάνια η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αυτή ένα πλωστάσιο στα χέρια της, έχει το εργαλείο το προενταξιακό, έχει την πολιτική CSDP, έχει ε, τη δική της πολιτική, έχει εσωτερικές πολιτικές και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα ε, για θέματα παρανομής διακίνησης όπλων, εμπορίας ανθρώπων και ούτω καθεξής. Με όλο αυτό λοιπόν το οπλοστάσιο είναι πολύ δύσκολο να επιτύχει κανείς τα αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και μερικές φορές αυτή η πολυμορφία των εργαλείων υπάρχει υποψία ότι είναι και η ε, ουσία του προβλήματος. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία, καλύτερη διακυβέρνηση ε, και αυτό όμως ε, μοιάζει όλοι να το λένε, δηλαδή ναι, καλύτερη στρατηγική προσέγγιση. Λέω όλοι. Εντάξει, όχι όλοι, ίσως να μην είναι απόλυτα αυτό, γιατί δεν θέλει κανείς να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το θέματα και μερικοί υποφελούνται από αυτή την κατάσταση και δεν θέλουν να βελτιωθεί, ε, τότε ακριβώς εξακολουθούν να ε, λειτουργούν τα πολλαπλά εργαλεία προς όφελος εκείνων που αντιδρούν. Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση, δύσκολο να αντιμετωπιστεί και αυτό που πρέπει να κάνουμε με τα περιφερειακά και τα εθνικά προγράμματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή που εκπροσωπώ, το που θέλουμε εμείς είναι να έχουμε μια πιο συντονισμένη προσέγγιση, μια περιφερειακή προσέγγιση αυτή των έξι κρατών της περιοχής να ενθαρρύνουμε ας πούμε τα δίκτυα των εισαγγελέων ή τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί όπως σας είπα επιθυμούμε να περάσουμε περισσότερο ε, στο ξέπλυμα του χρήματος γιατί Ας πούμε, μπορεί μία από αυτές τις χώρες να αποκτά χρήματα μέσα από το ξέπλυμα και μετά να τα επενδύει σε ακίνητη περιουσία στην γειτονική χώρα. Άρα δηλαδή χρειάζεται μία ε, πολυεθνική προσέγγιση. Ε, τα θέματα της αντιμετώπισης τρομοκρατίας δεν θα τα αφήξω γιατί είναι άλλη πιο κατάλληλοι. Όσον αφορά τις ε, θεσμικές αρμοδιότητες, ε, με αυτά τα θέματα ασχολείται περισσότερο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Δυστυχώς δεν έχουμε κανένα από αυτήν την υπηρεσία να είναι παρόντα εδώ. Θα πω και λίγα λόγια για τη μετανάστευση και μετά θα απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Τους τελευταίους έξι μήνες διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια νομιμοποίηση ε, της πολιτικής δύο κρατών που θίγονται, της ε, Φύρομ και της Σερβίας. Ένα είδος νομιμοποίησης ε, των παράτυπων ροών. Διευκόλυναν αν θέλετε τη διέλευσή τους από την Ελλάδα μέσω Φύρομ ε, μπορεί κανείς ε, να αποκτήσει πολύ εύκολα μία επιπρόσθετη υπηκότητα, αποκτά ένα χαρτί και μπορεί ε, για τρεις χώρες να διασχίσει μία χώρα και μετά για άλλες τρεις στη Σερβία. Και με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να αγοράσει εισιτήριο τρένου, να πάρει ταξί, να μπει σε λεωφορείο. Δηλαδή δεν είναι κανείς αναγκασμένος να απευθυνθεί στους διακινητές. Η νομιμοποίηση της διαδικασίας κατ' Δεν λειτουργήσε κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Όμως δεν βοήθησε στο να λυθούν όλα τα προβλήματα της ε, μεταναστευτικής κρίσης ε, ένα θέμα με το οποίο θα επιληφθεί αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως σας είπα με πολύ μεγάλη μου χαρά να απαντήσω σε ερωτήσεις από μέρους σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και εμείς ε, για όλα αυτά που ακούσαμε και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τις δικές μου τις ερωτήσεις, τις οποίες απευθύνω και στους δύο κυρίους ε, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρώτα απ' όλα θέλω να ρωτήσω το εξής. Μπορούμε κατά κάποιον τρόπο να περιγράψουμε την ε, ε, παράνομη εμπορία ανθρώπων, διακίνηση όπλων γιατί είναι σαφές ε, ότι αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη μεταναστευτική κρίση. Επίσης ε, δεν αποτελούν όλα αυτά καμία καινοτομία. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια και παλαιότερων ε, ενημερώσεων από επικεφαλής αποστολών, μας ε, ενημέρωσαν ότι εντοπίστηκαν ε, όπλα και πολύ σωστά αναφερθήκατε και στο, στην πορεία που οδηγεί στο Παρίσι. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ε, νομιμοποίησης των μεταναστών που διασχίζουν αυτές τις χώρες Μπορείτε κάπως ε, να εντοπίσετε από πού προέρχονται αυτοί οι μετανάστες, γιατί για μας, για την Υποπιτροπή Είναι πολύ σημαντικό για μας να μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση και να μπορούμε να εντοπίσουμε και τις επιπτώσεις που υπάρχουν στις ε, μεταναστευτικές ροές ή μάλλον από τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα σε μία από τις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής μας ακούσαμε ότι και πολλοί Αλγερινοί Φαίνεται ότι και αυτοί ακολούθησαν την διέλευση μέσα από τα Μαλκάνια, Βαλκάνια για να έλθουν στην Ευρώπη. Ισχύει αυτό ότι οι Αλγερινοί χρησιμοποιούν αυτή τη δυνατότητα. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο ε, στους ε, συναδέλφους. Ε, πρώτα απ' όλα έχει το λόγο ο κύριος Ράντος. Συγγνώμη, συγγνώμη, απαντάει η πρόεδρο. Ε, σε παρατήρηση του κ. Γκάλερ που δεν άκουσαν οι ήταν χωρίς μικρόφωνο. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. Ναι, θα είστε ο επόμενος. Κύριε Ράντο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Είπατε ότι 5-6 βαλκανικές χώρες συνεργάζονται ε, με την ε, Ευρώπη ε, και βεβαίως η αστυνομική συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να ανταλλαγούν πληροφορίες. Ε, αν και η συνεργασία κρατών μελών σε επίπεδο Europol δεν είναι αρκετά καλή και μάλιστα ένα μέρος ας πούμε της ευθύνης ε, πρέπει να φέρουν όσον αφορά τις πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι. και η συνεργασία ε, σε θέματα ε, προσφυγικών θεμάτων ε, σχετίζεται και με την επαφή που έχουν μεταξύ τους αυτές οι 5-6 βαλκανικές χώρες όσον αφορά τις αστυνομικές δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι αυτές οι χώρες βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο ένταξης και επομένως ρωτώ στα πλαίσια της ε, σταθεροποίησης των συμφωνιών σύνδεσης θα ήταν δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των έξι ε, ε, βαλκανικών χωρών όσον αφορά τις αστυνομικές δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ κύριε Μάικλ Γκράλερ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους ε, τους τρεις ε, εισηγητές. Ε, πραγματικά ακούσαμε πάρα πολλές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες που δεν τις ακούει κανείς κάθε μέρα. Και έχω μία ερώτηση προς τον κύριο Μπενεντέκ. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι Μέχρι τώρα η παροχή πληροφοριών από τα κράτη-μέλη προς τη Europol ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Γι' αυτό λοιπόν η Europol δεν μπορούσε να κάνει καλά τη δουλειά της ακριβώς γιατί δεν είχε στα χέρια της στοιχεία πληροφορίες για να έχει έτσι μια ολοκληρωμένη εικόνα. Ε, στη τελική ανάλυση ε, πρέπει κανείς να έχει μια γενική εικόνα και από αυτήν θα αποφεληθούν όλοι. Τώρα, λόγω του προσφυγικού μήπως άλλαξε η στάση των κρατών μελών, δηλαδή μήπως τώρα τα κρατημέλη δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν ξέρω, εγώ πολιτικά θεωρώ ότι και σε διμερείς επαφές όταν ένα κράτος μέλος ενημερώνει ένα άλλο ε, θα μπορούσε αυτή την πληροφορία να την κοινοποιεί ε, στο mail που στέλνει και προς την Europol έτσι ώστε και η Europol να αποκτά ε, τις απαραίτητες πληροφορίες. Έχουμε ένα παράδειγμα από τη Βαβαρία. Πριν από ένα μήνα η αστυνομία της Βαφαρίας είχε συλλάβει κάποιον που είχε παράνομα όπλα και στο GPS του είχε τελική, τελικός προορισμός Παρίσι. Ξέρετε τι έγινε, η Βαβαρία ενημέρωσε τις γαλλικές αρχές, αλλά είχε ξεχάσει να γράψει ότι πρόκειται για περίπτωση οργανωμένου εγκλήματος και επειδή υπάρχει πια αυτή, αυτός ο όγκος των πληροφοριών, ε, τι έγινε, δεν πρόσεξε κανείς αυτό το συγκεκριμένο mail και κάπου το θέμα χάθηκε. Αν όμως ε, είχε ενημερωθεί η Ευρωπόλ, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και θέλω να με ενημερώσετε τι γίνεται με όλα αυτά. Μία άλλη ερώτηση προς τον κύριο Τράουνερ. Εσείς ε, αναφέρατε το θέμα της ε, Βοσνίας Ερτσεκοβίνης, της Μπέρσκα, ο κύριος Ντόντικ θέλει να οργανώσει δημοψήφισμα το έχει κάνει πολλές φορές αυτό με διάφορα ερωτήματα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, ξέρετε κάτι, φοβάμαι μήπως αυτό το εκμεταλλευτεί ως πρόφαση να διατυπώσει το δημοψήφισμα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ενδεχομένως κάποιες ομοσπονδιακές αρχές του Σαράγεβο να μπορούν να έχουν αρμοδιότητα και για τη δική του την περιοχή. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι πολιτικά ε, πριν γίνει και πάλι αναφορά στον Dayton. Βέβαια, το Βελιγράδι δεν θα το κάνει αυτό. Το Βελιγράδι θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σω όμω βρεθεί κάποιο άλλο ενδιαφερόμενο. Ε, αυτό ήθελα να σα επισημάνω και ξέρετε γιατί. Για μην, να μην εκπλαγούμε αν και εκεί προκύψει άλλη αιστεία κρίση. Και μια άλλη ερώτηση. Είχατε πει ότι από τη Βοσνία και το Κοσοπέδιο έχουμε ξένους μαχητές οι οποίοι πάνε στη Συρία ίσως και από την Αλβανία και τη Μακεδονία, λέει ο μιλητής. Ε, υπάρχουν ε, και εκεί οι πολίτες που μετακινούνται προς τη Συρία. Θέλω λοιπόν να ξέρω, οι ξένοι μαχητές από τη Βοσνία, πώς είναι αναλογικά βέβαια αν τους συγκρίνουμε με αυτούς που πάνε από το Βέλγιο στη Συρία, ο αριθμός τους εν πάση περιπτώσει πρέπει να μας ανησυχεί, όχι. Ο κύριος Πίτσουλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις πανελίστες για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή τους που διεύρυναν τις προσωπικές μου γνώσεις όσον αφορά την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, κυρίως δε θέματα σχετιζόμενα με την ασφάλεια. Εγώ ε, ε, ε, έρχομαι από την Κροατία, είμαι μέλος και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και γνωρίζω αρκετά όσον αφορά την κατάσταση στο Κόσοβο και την Βοσνία Ζεχοβίνη. καλά είναι τα νέα τα οποία αναφέρατε στην παρουσίασή σας όσον αφορά την προώθηση της ε, ε, διείσδυσης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στα Δυτικά ε, Βαλκάνια και ότι προχωρούν διάφορες διαδικασίες σύνδεσης ε, με, το, ε, με τη Σερβία και με το Μαυροβούνιο. Αυτά είναι πολύ καλά νέα γιατί όσο προοδεύουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων βελτιώνεται η κατάσταση σε μια αποσταθεροποιημένη γενικά περιοχή. Ε, μην λησμονείτε ότι η προσφυγική κρίση ε, έχει ε, ξεκινήσει στην περιοχή εκεί και πρέπει να πω ότι η κρίση ξεκίνησε μεταξύ δύο χωρών, όχι μόνο μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και μελών Σέγγεν, Ουγγαρίας και ε, Ελλάδος. Εκεί ξεκίνησαν, ας πούμε, ε, να συμπεριφέρονται οι χώρες διαφορετικά ε, και με άλλα πρότυπα, υψώνοντας φράχτες και αυτό προκάλεσε την αλλαγή διαδρομής των ε, προσφύγων ε, προς την Φύρομ ε, και λοιπά. Επίσης, πρόκειται ε, ε, ε, επίσης ταυτόχρονα με την ροή την προσφυγική έχουμε και μία σειρά αλλαγών και μία σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Τουρκία, Ελλάδα και σιγά σιγά και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αυτό ταυτίζεται ε, ε, συγκυριακά τουλάχιστον ε, με την προσφυγική κρίση καθώς επίσης και με την ιδιαίτερα ηλυπή οικονομική διάρθρωση πολλών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Βέβαια η κατάσταση μπορεί να αλλάξει εν μία νυχτή. Ερώτηση λοιπόν, πώς προβλέπετε τις εξελίξεις σε περίπτωση όπου η Γερμανία, η Αυστρία και ίσως και άλλες χώρες αλλάξουν την πολιτική τους ε, τοποθέτηση χωρίς να λαμβάνουν ε, υπόψη ε, την κατάσταση στα Δυτικά Βαλκάνια, αρχίσουν επομένως ε, να αντιμετωπίζουν με τρόπο εντελώς διαφορετικό τους άτυπους μετανάστες. Πώς βλέπετε την κατάσταση, πώς μπορείτε να, πώς, μπορείτε να φανταστείτε ότι θα εξελιχθεί η κατάσταση και να μου πείτε α, β, γ, αυτό θα συμβεί εάν και εφόσον εξελιχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα ε, να δώσω στους έγκριτους καλεσμένους μας ε, τον λόγο για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας και επομένως ε, να απαντήσουν σε κάποια από τα ερωτήματά σας και ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει και ένας δεύτερος γύρος ερωτήσεων εάν κάποια σημεία παραμείνουν ασαφή. Κύριε Καθηγητά, Thank you for the uh, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μερικές από αυτές. Όσον αφορά την ε, ε, αστυνομική συνεργασία της περιοχής, βεβαίως αυτή ε, καλλιεργείται και, από την, και, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην υπάρξει μόνο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αστυνομικών αρχών αυτών των χωρών, αλλά και συνεργασία μεταξύ τους. Ε, υπάρχει μια σχετική οργάνωση η οποία ε, δρεύει στην ε, Σόφια και η οποία συντονίζει ας πούμε αυτήν την συνεργασία καθώς επίσης και, την, και κάποιες διεργασίες επιβολής του νόμου. Ε, πρόκειται για μια συμφωνία η οποία βασίζεται στην συμφωνία Σέγγεν, δηλαδή παρουσιάζει κάποια ίδια ε, χαρακτηριστικά και προωθεί και την ε, διακρατική συνεργασία. Επίσης, ε, πραγματικά θα πρέπει να παρακολουθούν ε, οι πολιτικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης από, την, από κοντά την ε, κατάσταση. καταλαβαίνουμε ότι οι πολίτες γενικά δίνουν, αποδίδουν μεγάλη προσοχή και σημασία στους κοινωνικούς ε, στα κοινωνικά προβλήματα, στα οικονομικά προβλήματα. Τα εθνικιστικά ίσως έχουν περάσει πλέον ε, σε δεύτερη ε, μοίρα και επομένως και σε αυτά τα δημοψηφίσματα τα οποία έχουν αναφερθεί ε, κατά του ΝΑΤΟ ε, ε, έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, έχουν παριθέσει διάφοροι φορείς. Το Βελιγράδι τώρα, για να αναφερθώ στο άλλο θέμα που θίξατε, συνεργάζεται στενά με τις αρχές της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και επομένως δεν φαίνεται ε, να στηρίζει υπερβολικά ή ε, ιδιαίτερα την πρωτοβουλία για δημοψήφισμα της Ρεπούμπλικας Έψκα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, ε, κ. Πενέντε. Να ξεκινήσω με τις δικές σας ερωτήσεις, κυρία Πρόεδρε, για το αν σχετίζεται το αθρεμπόριο όπλων με την προσφυγική κρίση. Αυτό που βλέπουμε με την αξιολόγηση ε, σοβαρής εγκληματικής απειλής ε, που δημοσιεύει η Ευρωπόλ είναι ότι έχουμε εξειδίκευση ε, και πηγαίνουν στις πιο αποδοτικές κερδοφόρες αγορές οι εγκληματικές ομάδες. Βέβαια η διευκόλυνση της παράτυπης μετανάστευσης ήταν θετική για αυτό το εμπόριο και επομένως αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι τα πιο επαγγελματικά εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων και σε ό,τι αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία, το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι ορισμένα από τα όπλα που χρησιμοποιούν οργανωμένε εγκληματικέ ομάδε στην Ένωση τα έχουν φέρει από τα Δυτικά ε, Βαλκάνια ε, με λαθρεμπόριο, γιατί μπορεί κανεί να τα ε, ανοιχνεύσει και έχουμε στοιχεία ότι προέρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια και σε ό,τι αφορά τις πρόδρομες ουσίες έχουμε σχέσεις με τα οπλοστάσια που υπάρχουν στα Δυτικά Βαλκάνια και τις εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έχουμε, τέτοια στοιχεία. Ο κύριος Σοράτζ, ο κύριος Γκάλερ, συμφωνώ μαζί σας ότι τα κράτη-μέλη και η Europol δεν συνεργάστηκαν επαρκώς. Το έδειξαν και οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις. Παρότι υπήρχαν τα μέσα και ανταλλαγή ε, πληροφοριών ε, ήταν δυνατή, θα μπορούσε με αυτή την ανταλλαγή που είναι ασφαλής ε, όλα τα κράτη-μέλη να είχαν δώσει πολύτιμες πληροφορίες στους ομολόγους τους. Δεν έγινε όμως στον αναμενόμενο βαθμό. Έχω εδώ κάποια στοιχεία για παράδειγμα, άρθρο 36 προειδοποίησης, ο σύστημα πληροφοριών. Χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα από λίγα κράτη-μέλη μόνο. Με αυτή τη δυνατότητα οι πήκοοι τρίτων χωρών θα μπορούσαν να είχαν ε, ταυτοποιηθεί ω υποτέλεση ε, τρομοκρατικών ενεργειών. Επίσης, δεν είχαμε στοιχεία στο σύστημα της Ευρωπόλ αν το είχαν αυτά τα στοιχεία ε, μετά το Παρίσι, θα είχαν πάρει οι Βέλγοι, οι Γάλλοι συνοριοφύλακε από τους Βέλγους συνοριοφύλακε ή ε, Τούμπαλιν τα στοιχεία και θα είχαν ε, σταματήσει στα σύνορα αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, μπορούμε να έχουμε βελτίωση, μπορούμε να βελτιώσουμε από μόνοι μας τα πράγματα, τεχνικά μέσα όμω υπάρχουν. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει 25 Ιανουαρίου ένα Ευρωπαϊκό Τμήμα Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας ε, στο πλαίσιο της Ευρωπόλ. Έχουμε επιχειρησιακά καθήκοντα που πρέπει να επιτελούμε για να αντιμετωπίζουμε τις τρομοκρατικές απειλές, αλλά υπάρχει και το σκέλος της ανταλλαγής πληροφοριών πλέον, που αυτό έλειπε, το είδαμε στις τελευταίες ε, επιθέσεις, στο Παρίσι συγκεκριμένα. Κάτι άλλο που θέλω να πω αφορούσε την ε, αστυνομική συνεργασία. Υπάρχει σύμβαση για την Ιταλική Ευρώπη, τον έφερε ο Φλόριαν για την αστυνομική συνεργασία. Ένα πρόσφατο παράδειγμα, ε, το έχουμε επεξεργαστεί ο Άντριου και εγώ, είναι ένα ειδικό μέτρο που ενέκρινε για την Φύρον πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δίνει τη δυνατότητα σε διάφορα κράτη-μέλη να στέλνουν ε, συνοριοφύλακες στη Φύρον ως προσκεκλημένους των εισαγωγικών για να ελέγχουν τα σύνορα με την Ελλάδα. Κάποιες χώρες έστειλαν συνοριοφύλακες στην Μακεδονία με βάση αυτή τη σύμβαση ε, αστυνομικής συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χρησιμοποίησαν δηλαδή αυτό το περιφερειακό πλαίσιο για μια πολύ ευαίσθητη, πολύ λεπτή αποστολή, γιατί στέλνουν δικούς τους συνοριοφύλακες. Άρα, κατά το μακεδονικό δίκαιο και με μακεδονική διοίκηση και πηγαίνουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, να διαχειριστούν σύνορα μεθόρα με την Ελλάδα. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομικό μέσο. Εμείς βέβαια εδώ και χρόνια έχουμε εκφράσει την προτίμησή μας για στενότερες σχέσεις των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπόλη. Από ε, θεσμικής πλευράς λοιπόν αυτή είναι η προτίμησή μας και αυτή είναι η συμβολή μας προς αυτές, η συμβούλή μας προς αυτές τις χώρες. Να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά περιφερειακά βήματα ε, για την αστυνομική συνεργασία. Rasmus. Ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω. Κυρία Πρόεδρε, εσείς είπατε ότι υπάρχουν μη Σύριοι, μη Ιρακινοί, μη Αφγανοί που όμως ε, προσποιούνται ότι είναι. Και αυτό σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και υπάρχουν δύο-τρεις παράγοντες για Αλγερινούς και Μαροκινούς ε, ακούμε ε, συνήθως. Οι Μαροκινοί μπορούν να μπουν εύκολα στην Τουρκία χωρίς να χρειάζονται βίζα. Άρα και μετά μπορούν να προσποιηθούν πολύ εύκολα ότι είναι Σύριοι ή Ιρακινοί ή Αφγανοί όταν φτάνουν στα ελληνικά νησιά. Και όταν φτάσουν εκεί και αν πείσουν ε, αυτούς που τους παίρνουν συνέντευξη και είναι σχετικά εύκολο να τους πείσουν γιατί μέχρι τώρα η έλεγχη δεν ήταν όσο αυστηρή θα θέλαμε. Από ό,τι φαίνεται και με την υποστήριξη που δούμε στην Ελλάδα, το είπε και ο Μάρτιν, κάπως βελτιώνται τα πράγματα, άρα πέρασαν πολύ. Εγώ πήγα πιο πολύ στη Φιρόμ βέβαια και είδα τη δική τους εμπειρία ε, στη Μεθόριο που έχουν με την Ελλάδα τι μας λένε, ότι αυτοί που έρχονται με αυτά τα ελληνικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα νησιά, Πρώτον, με την πρώτη ματιά το 89% βλέπουν ότι είναι πλαστό το έγγραφο που έχουν και δεύτερον δεν έχουν την ε, εθνικότητα που λένε ότι έχουν, είναι σαφές, στο 80-90% των περιπτώσεων. Εσείς είπατε ενίσχυση πολλών κρατών και ε, από τη Σερβία και τη Φύρο να βοηθήσουν την ε, διαχείριση της Νότιας ε, Μεθορίου και από το Δεκέμβριο. Νομίζω η Κροατία έστειλε ήδη το Δεκέμβριο μια μικρή ομάδα ανθρώπων και ακολουθούν και άλλες χώρες όπως είπα και η Σερβία. Η νομική βάση είναι ή η πολυμερή σύμβαση, PCC ή διμερή συμφωνία. Τα είπατε και εσείς. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς είπαμε ότι θα υποστηρίξουμε, ε, παραδείγματος τη ε, αναλαμβάνοντας μέρος του κόστους. Έχουμε τους μισθούς, τα οχήματα, τον εξοπλισμό, τις μερίσχες αποζημίωσεις, αλλά η διαμονή, η διατροφή και τη βενζίνη πληρώνεται από τη Μακεδονία. Είναι μακεδονική αποστολή, αλλά δέχεται υποστήριξη στα άλλα που σας είπα, λόγω της νομικής αυτής βάσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί μέσω του ΙΠΕΡ. Και με τις περιπολίες θέλουμε να έχουμε βελτίωση. Αλλά θέλουμε να ενισχύσουμε την ικανότητα και τη δυνατότητα με βιομετρική δυνατότητα καταγραφής, ε, να βελτιώσουμε την καταχώρηση, να καταγράφονται όσοι παίρνουν τα σύνορα με πολύ πιο σοβαρό τρόπο. Και μετά να υπάρχει διασύνδεση με τη βάση δεδομένων των Σκοπίων. Όχι άμεσα δυστυχώς με την βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερη η γνώση που θα, θα ξέρουν ποιος έχει περάσει. Θα μπορούμε να εντοπίζουμε, να ταυτοποιούμε πολύ πιο εύκολα αυτούς περνάνε Γιατί ουσιαστικά μέχρι στιγμής έχουμε τις ε, δηλώσεις των ίδιων των ανθρώπων. Και δακτυλικά αποτυπώματα, βιομετρικά, ναι, τις επόμενες εβδομάδες. Και συνεργαζόμαστε με τον IOM, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ε, τώρα, σχέδιο Α, σχέδιο Β, σχέδιο Γ. Σχέδιο Γ δεν ξέρω. Αλλά για σχέδιο Α, σχέδιο Β έχει γίνει πολλή συζήτηση και νομίζω ότι πιο πολύ το θέμα είναι το πότε θα χρειαστεί ένα τέτοιο σχέδιο και όχι αν. Παραμένουν πολύ ψηλοί αριθμοί των διελεύσεων, 2.000 τη μέρα από τις αρχές του έτους και που είναι και οι πιο άσχημες καιρικέ συνθήκες και πιο μεγάλη κίνδυνη για τη διέλευση διαθαλάσσης. Άρα, ίσως στάσουμε στα, στους αριθμούς του φθινοπόρου της περσινής χρονιάς. Δεν έχει αλλάξει. Πολλοί θέλουν να περάσουν ε, διαθαλάσσια από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη, Γερμανία, Αυστρία, ε, θα δούμε τι θα κάνουν. Ό,τι γίνεται όμως downstream, κατάντι, μέχρι και κλείσιμο συνόρων, έχουν α, ε, αμέσως επιπτώσει και προς τα πάνω. Αν κλείσει ε, η Σερβοκρατική Μεθόριος, θα κλείσει μετά και η Μακεδονία τα σύνορα, θα κλείσει μετά ε, τα σύνορα με την Ελλάδα και ήδη βλέπουμε περιορισμούς σε αυτή τη διαδρομή. Το φθινόπωρο πέρυσι κατά εθνικότητες, αλλά έγινε συντονισμένα με όλες τις χώρες ταυτόχρονα. Αν υπάρξει κλείσιμο συνόρων θα γίνει γρήγορα. Τώρα, αναμφίβολα κάποιοι θα παγιδευτούν Στι χώρε. Ιδίω εδώ μιλώ για Φιρούμ και Σερβία. Και τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μπορούμε να εικάσουμε το ότι μπορεί είτε να μείνουν εκεί περιμένοντας να μετεγκατασταθούν, είτε θα πέσουν στα νύχια των διακινητών. Θα τους δουν ως ε, ε, ευκαιρία για κέρδος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αυξήσουμε τη δυνατότητα υποδοχής των χωρών της περιοχής και κατά μήκο όλη αυτή τη διαδρομή, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να φιλοξενηθούν με ξοπρεπείς συνθήκε και θέλουμε να ε, να πραγματοποιήσουμε τέτοια project στην περιοχή. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, αναφέρθηκαν ήδη τα περισσότερα στοιχεία, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο αφορά την Ελλάδα. Η Ελλάδα ε, μάλλον να το πω διαφορετικά, το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό που θα γίνει αύριο θα προσπαθήσει να λύσει ορισμένα από τα ζητήματα τα οποία εδώ και μήνες αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Ε, μία από τις ε, ε, διαφορετικές ε, που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την, ε, την κατανομή των προσφύγων είναι το πρόβλημα της επιστροφής στην Ελλάδα βάσει του συστήματος του Δουβλίνου. Επίσης υπάρχουν ζητήματα ανθρωπίνων ε, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά τους ετούντες άσυλο στην Ελλάδα. Ε, ε, ελπίζω ότι η Ελλάδα λιγότερο, σύντομα, συντομότερα θα μπορέσει να ενταχθεί πραγματικά στο σύστημα του Δουβλίνου. Θα υπάρξουν τα hot spots σωστά και λειτουργούντα Έχουμε περισσότερα προβλήματα στην Ελλάδα από ό,τι στην Ιταλία. Σχόλια εκτό μικροφώνου δεν ακούν οι διερμηνείς. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν δύο. Αλλά από ό,τι φαίνεται ε, η πρόθεση είναι να ξεκινήσει, να ανοίξει ένα hot spot σε κάθε νησί και η ιδέα είναι ότι όταν ε, θα έχουν ολοκληρωθεί τα hot spots, όταν η Ελλάδα θα είναι ξανά στο σύστημα Δουβλίνου, όταν θα λειτουργούν κανονικά τα σύνορα μεταξύ Φύρων Ελλάδας ε, και επομένως και η Frontex θα βοηθάει έτσι ώστε να υπάρχουν οι σωστές έξοδοι από την ε, Ελλάδα τότε από την μακεδονική πλευρά, λέει ο μιλητής, ε, θα ε, ε, λειτουργήσουν καλύτερα και τα σύνορα από εκεί. Είναι ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πρέπει υποχρεωτικά να μπουν στο σύστημα επανεγκατάστασης. Ε, υπάρχει και το ζήτημα ε, των περιπτώσεων περιπτώσεις αυτές, ε, άνθρωποι οι οποίοι προωθούνται προς χώρες που δεν είναι η επιλογή τους, τότε βγαίνουν, αποσύρουν το αίτημα για άσυλο έτσι ώστε να ξαναμπούν στο σύστημα με καινούργιες διαδικασίες. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε αυτά τα hot spots στην Ελλάδα, να βεβαιώσουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να μπει στο σύστημα Δουβλίνου, ότι θα γίνονται οι σωστή κατάλληλη έλεγχη μεταξύ, σύνορα μεταξύ Ελλάδας ε, και ε, Φύρων, έτσι ώστε οι άνθρωποι υποχρεωτικά να μπαίνουν στο σύστημα επανεγκατάστασης. Λοιπόν, επειδή έχουμε χρόνο, ε, να κάνω κι εγώ δύο ερωτήσεις και θέλω, αν θέλουν, να θέλουν τους συναντέλφους να κάνουν και εκείνοι το ίδιο. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, δυστυχώς. κοιτάξτε, αυτούς τους ε, ξένους μαχητές στη Βοσνία που ρωτήσατε. Πριν απαντήσω να σας πω κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει για τη Europol και για το Κωσυφοπαίδιο. Γιατί είπατε ότι το Κωσυφοπαίδιο είναι η μόνη χώρα η οποία δεν έχει υπογράψει ακόμα συμφωνία συνεργασίας με τη Europol. Να σας πω όμως ότι οι πληροφορίες διοχετεύονται μέσω της Eulex και υπάρχει ένα κράτος στη Σουηδία που έχει προσφερθεί να παίρνει αυτές τις πληροφορίες ε, ε, και να τις στέλνει ε, στην Europol. Αλλά πράγματι δεν υπάρχει επίσημη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε Europol και 25 και αυτό είναι ένα θέμα για την ασφάλεια της περιοχής. Και εδώ επιτρέψτε μου μία υποσημείωση δική μου σχετικά με το θέμα που ρωτήσατε για τους ε, τζιχαντιστές ε, στα Βαλκάνια. Ρωτήσε τον αριθμό. Κοιτάξτε, στη Βοσνία είναι οι περισσότεροι. 340. Μετά έρχεται το 25 η Μακεδονία σε καμιά ε, Κοσαριά είναι εκεί. Περιορισμένοι αριθμοί και για την Αλβανία, Σερβία περισσότεροι. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Βοσνία βρίσκεται ε, σε αυτό που ισχύει και στη Δυτική Ευρώπη, Βέλγιο, Γαλλία, εδώ είναι οι περισσότεροι τζιχαντιστές. Το θέμα είναι ότι στη Βοσνία υπάρχει τέτοια κατακαιρματισμένη δομή, δεν υπάρχει συνεργασία, ως εκ τούτου ε, εκεί πράγματι υπάρχει μεγάλο θέμα ασφάλειας. Ναι, κατά κάποιον τρόπο ακολουθεί η Βοσνία της εξελίξεις που υπάρχουν και στη Δυτική Ευρώπη, όμως επειδή υπάρχει άλλη υποδομή, υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι στα δυτικά κράτη. Η πρόεδρος, η δική μου η πρώτη ερώτηση έχει σχέση περισσότερο με το επόμενο θέμα της μερικής διάταξης που είναι η ενημέρωση για τη UNAFOR, ε, αποστολή ενημέρωσης. Αναφέρεται κάποιες αλλαγές ε, στις ε, μεταναστευτικές δομές ε, στα Δυτικά Βαλκάνια μετά την ανάπτυξη της UNAFOR στη Σόφια. Και τι ακριβώς περιμένετε Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ανανεωθεί η εντολή της UNAFOR έτσι ώστε να ακολουθήσει η δεύτερη ή έστω και η τρίτη φάση που να αφορά ε, στα εδάφη της ε, Λιβύης και τα χωρικά της Ήδατα. Ε, και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά περισσότερο ε, σε, στη βιντεο conference του κύριου Τσίγκαν, στο ρόλο της Τουρκίας. Κάπως το θίξατε, ακροθυγός όμως, εγώ θα ήθελα ε, κάποια ε, εμβάθυνση σε αυτό το θέμα και από τους τρεις ε, εισηγητές. Και ο κύριος Πρόντι έχει το λόγο. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ από την αρχή της ε, συνάντησης, αλλά θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπενεντίκτ, γιατί έθιξε το θέμα των hot spots. Στην ομιλία του. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το εξής. Αυτά τα hot spots τι είναι αυτά. Ποιος τα αποφασίζει, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει. Θα είναι δηλαδή ένα είδος ε, διεθνούς ε, προσωπικού ε, που θα επαντρώσει αυτά τα hot spot. Θα είναι μόνο Έλληνες, τι θα είναι. Δεν ξέρω. Ποιο είναι το σχέδιο για τα hot spot, γιατί μιλάμε για τα hot spot, δεν ξέρω τώρα, περίπου κάνα χρόνο νομίζω <coughs> και δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ούτε ένα. Ωραία, λέει η πρόεδρος. Ε, δεν θέλει κανείς άλλος από την βλέπω να κάνει ερώτηση. Ε, μπορείτε παρακαλώ να λάβετε το λόγο, οι εισηγητές. Λοιπόν, ε, να δούμε λιγάκι το ρόλο της Τουρκίας. Αν διαβάσει κανείς ε, την τελευταία έκθεση ε, εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αποκομίσει κανείς την άποψη ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωση, αλλά δεν είναι τόσο κολλή όσο ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η Τουρκία έκανε κάποια βήματα, άνοιξε την αγορά εργασίας για τους πρόσφυγες, προσπάθησε να εντάξει κάποιους πρόσφυγες στα σχολεία, Άρα δηλαδή τα κίνητρά τους να έρθουν στην Ευρώπη περιορίζονται. Επίσης η Τουρκία προτίθεται να θεσπίσει κανόνες για να εναρμονιστεί με την ομοθεσία που υπάρχει σε εμά για την προστασία των δεδομένων. Θέλει επίση να συνεργαστεί περισσότερο για θέματα ασφάλειας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήλπιζε περισσότερα να περιστεί ο αριθμός των προσφύγων. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όσο ήλπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία ε, παίζει σε πολλά παιδεία, σε πολλά γήπεδα. Η Τουρκία θέλει να ενισχυθεί περαιτέρω έναντι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και το θέμα το μεταναστευτικό βολεύει την ε, τουρκική κυβέρνηση. Άρα δηλαδή ε, τίθεται το θέμα μήπως ε, τελικά η Τουρκία δεν έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει ουσιαστικά το μεταναστευτικό. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας από τη δική σας την ερώτηση, κυρία Πρόεδρος, Θέλω να σου πω, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονα τη UNAFOR αλλά εφόσον μιλάμε για την Τουρκία που είναι το άλλο σκέλος της εξίσωσης και θα συζητηθεί αύριο αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο ε, μου έχει επαφές με τους Τούρκους και αυτό που έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί ε, το σχέδιο που έχει καταρτιστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα μεγάλο σκέλος αυτού αφορά την, ε, το να μην έρχονται πρόσφυγες από την Τουρκία ε, στα ελληνικά νησιά. Το ε, συζητείται σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Είναι όμως θέμα κλειδί. Αν θέλει κανείς να περιορίσει τις ε, ροές ε, από την Τουρκία, το Λίβανο και την Ιουρδανία, πρέπει κανείς οπωσδήποτε να μιλάει με την Τουρκία. Ε, τώρα, σχετικά με τις προσδοκίες δεν είμαι τόσο αισιόδοξο όσο θα έπρεπε να είμαι βλέποντας τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία. Τώρα δεν βλέπω να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Δεν διαφαίνονται στον ορίζοντα. Πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας, άρα δηλαδή η συνεργασία με την Τουρκία είναι απολύτω απαραίτητη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Τουρκίας. Επίσης ό,τι αφορά την Ελλάδα και αυτά να πάνε καλά και όλες οι άλλες χώρες ε, στα Δυτικά Βαλκάνια να τηρήσουν τις ε, δεσμεύσεις τους του Οκτωβρίου. Και αυτό θα εμποδίζει τους ανθρώπους να φεύγουν ε, θα μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τις μεταναστευτικές ροές. Πρόβλημα. Ο καιρός. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων. Μετά αν υπάρχει και άλλη πιο έντονη σύγκρουση στο Χαλέπι και εκεί... Ε, και αυτό θα επηρεάσει. Πολλοί έρχονται όχι από τη Συρία, αλλά από τους καταβλισμούς και ξέρουμε από την Ιορδανία, το Λίβανο και την Τουρκία ότι φιλοξενούν ε, πάρα πολλούς. Ένα άλλο θέμα λοιπόν είναι να ε, βελτιωθούν οι συνθήκες ε, στην Τουρκία έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν τόσα κίνητρα για να φύγουν. Όσον αφορά την ερώτηση για τα hot spot, θα είναι υπό ελληνική διοίκηση, αλλά βέβαια με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Frontex. Ο ρόλος τους είναι να ε, ταυτοποιούν και να καταγράφουν τους νεοαφιχθέντες. Υπάρχει τελευταία δήλωση της Επιτροπής της 12 η Φεβρουαρίου. Εκεί μπορείτε να ανατρέξετε και να την βρείτε στο, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτή είναι η πρόταση προς το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Ένας από τους αριθμούς που αναφέρεται λέει ότι όσοι ε, δακτυλοσκοπούνται από το 8% του Σεπτεμβρίου αυξήθηκε στο 55% το Δεκέμβρη και στην Ιταλία από 36% σε 67%. Αυτά όλα με βάση ε, τη λειτουργία των hotspot. Έχουμε λοιπόν πολλούς εμπειρογνώμονες που μπορούν να δίνουν καλές συμβουλές και στους Έλληνες και στους Ιταλούς για το πώς να καταγράφουν τους νεοαφιχθέντες, τους παίρνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα, αυτά πάνε στη Eurodac και αυτό θα καθορίσει ε, τα μελλοντικά βήματα ε, μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ε, να μπορούν αυτοί να μπουν στο μηχανισμό επανεγκατάστασης, να μπορούν να επανεγκατασταθούν στη Λετωνία ή στη Φινλανδία. Τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και αυτό θα συζητήσει αύριο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κύριος Ράσπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα της Τουρκίας, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η Τουρκία είναι καθοριστική και πράγματι πρέπει να το πούμε ότι οι Τούρκοι, να το αναγνωρίσουμε αυτό, ότι έχουν δεχτεί ένα τεράστιο αριθμό προσφύγων και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι το υπαριθμό ένα. Το δύο είναι ότι είναι σκληροί παίκτε. Διάβασα πρόσφατα ε, τα πρακτικά της συνάντησης ε, Τούσκ ε, και Γιούνκερ με τον πρόεδρο της ε, Τουρκίας. Δεν ξέρω τότε αν ήταν πρόεδρος υπουργός, τέλος πάντων πρόεδρος ήταν όταν συναντήθηκαν. Ήταν ήδη πρόεδρος. Μπας περιπτώσει το θέμα είναι ότι ε, είναι πολύ σκληροί παίκτες και από τη Γενική Διεύθυνση της ε, Διεύνησης ε, έχουμε πολλές επιφυλάξεις για την αντιμετώπιση των δημοσιογράφων, την ελευθερία του τύπου και πολλά παρεμφερή. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει κανείς να γνωρίσει ότι όταν έχει να κάνει με την Τουρκία έχει να κάνει με μια χώρα ε, που έχει ένα τεράστιο δυναμικό. Αν θέλουν μπορούν να τους διώξουν αυτούς που βρίσκονται και αν θέλουν μπορούν να τους κρατήσουν. Και ένα από τα βασικά μηνύματα είναι ότι αυτό που απασχολεί περισσότερο είναι τα θέματα της ε, ακτοφυλακής. Ενώ θα έπρεπε κανείς, αντί να ασχολείται με αυτούς που φεύγουν στη θάλασσα, το τι γίνεται μέσα στην ίδια τη χώρα, την Τουρκία, πώς αντιμετωπίζονται οι διακινητές και πολλά. Αυτό είναι περισσότερο θέμα χωροφυλακής και όχι τόσο ακτοφυλακής. Και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με το Συριακό. Ε, αυτή τη στιγμή οι μισοί έρχονται από τη Συρία. Το 40% και περίπου το 55% από το, τις άλλες δύο χώρες, το Ιράκ και το Αφγανιστάν και λίγοι ακόμα οι οποίοι έχουν κάποιο άλλο διαβατήριο που δεν το αναφέρουν καν. Άρα δηλαδή ακόμα και αν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Συρίας, θα εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα προσφύγων. Τώρα ε, υπάρχει αυτή η δίωδος μέσα από την ε, Τουρκία η οποία μοιάζει να λειτουργεί και άρα εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας για την οποία πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ενημερώσατε. Φυσικά η Επιτροπή μας εστιάζει κυρίως ε, στην ασφάλεια και στην άμυνα. Γι' αυτό και προσπαθούμε να στρέφουμε τις ερωτήσεις μας γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ήταν πάντως πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση που μας κάνατε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.

be Ευχαριστώ πολύ. Ξανακαθίστε παρακαλώ. is of... Uh, Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Θα ασχοληθούμε με κάτι το οποίο συνέβη πρόσφατα, ε, δηλαδή την αποστολή ενημέρωσης ε, στην ε, Σόφια. στη Ρώμη, συγγνώμη, τον Φεβρουάριο ε, σχετικά με ενημέρωση για την Euronav4 στην ε, Σόφια. Ε, είχαμε τον κύριο Λορέντσο Τσέζα από την Ιταλία. Τα οργάνωσε όλα πολύ καλά. Ήρθαμε σε επαφή με εκπροσώπους της Ιταλικής Κυβερνήσεως, καθώς επίσης και με εκπροσώπους ε, του Κοινοβουλίου, τον, ε, καθώς επίσης και με εκπροσώπους ε, think tanks. Εγώ ήμουν επικεφαλής της αποστολής και ε, όταν έφυγα εγώ γιατί έπρεπε να πάω στην Κρήτη, ο κύριος Καστανάλος πήρε το, την θέση μου. Και είχαμε και τον κύριο Τσέζαμ, την κυρία Άννα Γκόμες, την κυρία Γιάλα Σέντερ και τον κύριο Χαβιερνάτ. Την πρώτη ημέρα της επίσκεψής μας, είχαμε ε, την ενημέρωση από πλευράς των ε, υπουργών και πρωθυπουργών που είναι υπεύθυνοι για τα ευρωπαϊκά ζητήματα και είχαμε την ευκαιρία να θίξουμε σειρά ε, θεμάτων, όχι μόνο για θέματα ασφάλειας, αλλά και για άλλα ζητήματα, κυρίως για την προσφυγική κρίση και όλα τα με αυτήν σχετιζόμενα θέματα. Είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε ε, τις ε, ε, απόψεις της τελικής δημοκρατίας για το θέμα αυτό. Η επόμενη μέρα, σχεδόν εξ ολοκλήρου, αφιερώθηκε στην επίσκεψη των, ε, ε, του κέντρου της ε, UNAV4. συναντήσαμε λοιπόν όλα τα μέλη, τα υψηλόβαθμα της αποστολής. Είχαμε μία εκτεταμένη επομένως ενημέρωση και ο Ναύρος Κρεντεντίνο δεν ήταν διαθέσιμος ακριβώς εκείνη τη στιγμή, αλλά βεβαίως ε, είχαμε την ε, καλύτερη δυνατή ενημέρωση από τον ε, αντικαταστάτη του και ο Ναύροχος μας υπεσχέθη ότι στις επερχόμενες ακροάσεις θα είναι μαζί μας Uh, route for, for exchange. Και θα έχουμε την, την ευκαιρία λοιπόν να ανταλλάξουμε απόψεις και μαζί του. Επίσης, συναντήσαμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Αλφάνο, ο οποίος μας έδωσε μία ευρυτάτη έποψη και επισκόπηση όλων των θεμάτων ε, ε, που σχετίζονται με την προσφυγική κρίση και το πώς την αντιμετωπίζει η Ιταλία. Επίσης είχαμε και τον αναπληρωτή ε, Υπουργό Άμυνα, ο οποίος μας έδωσε τη δικιά του επισκόπηση. Σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ιταλία το θέμα. Εγώ προσωπικά θεώρησα ότι αυτή η επίσκεψη ήταν εξαιρετικά επιμορφωτική, ιδιαίτερος σημαντική και με την επίσκεψη αυτή στην ε, e Nav Format Sofia ε, είχαμε την ε, δυνατότητα να δούμε ποιες είναι οι καθημερινές δραστηριότητες της ε, ε, EU for Med Sofia ε, και είδαμε και τον τρόπο με τον αντιμετωπίζουν την κατάσταση σε καθημερινή βάση. Και είδαμε και πώς σε πραγματικό χρόνο αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και γιατί πρόκειται για μια εμβληματική ε, διαδικασία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί ε, και πραγματικά ήταν μια ιδιαίτερος ευχάριστη η αποστολή αυτή. Μήπως θέλει η κυρία Γιάλα Σέντερ να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ε, θα ήθελα ε, και εγώ να σας εκφέρω τη δικιά μου ε, άποψη, βεβαίως λέγοντας ότι συμφωνώ απολύτως με την άποψη που δώσατε εσείς, ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η αποστολή και επίσης σημαντική λόγω του έυρους των πληροφοριών που είχαμε και την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης και όσον αφορά τα εσωτερικά ζητήματα και όσον αφορά ε, την ε, άμυνα και σε αυτή τη συνάντηση που είχαμε τη δεύτερη μέρα. Ε, είχαμε από πρώτο χέρι λοιπόν πληροφόρηση για μία αποστολή ε, η οποία είναι παρόμοια κατά κάποιο τρόπο με την επιχείρηση Αταλάντη ε, και ε, πρόκειται για μια επιχείρηση στην θάλασσα της Μεσογείου με όλα αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία και τα στοιχεία επιπλοκής λόγω και των γειτονικών χωρών αλλά διαπιστώσαμε ότι στην παρούσα φάση τα πράγματα είναι θετικά δηλαδή ότι έχει έχουν επιτευχθεί οι δύο εντολές, αυτό δηλαδή της διάσωσης ζωών. Ε, ε, πολλές ζωές έχουν σώσει σε αυτή τη δεύτερη φάση, αλλά ε, κατάφεραν επίσης να ε, ε, καταστρέψουν τις βάρκες των ε, διακινητών που ήταν ακριβώς το δεύτερο σκέλος της εντολής τους καθώς επίσης και όσον αφορά την συλλογή πληροφοριών και στην ανταλλαγή πληροφοριών με την Ιταλική κυβέρνηση. Ε, αλλά και με τον εκπρόσωπο του ε, επικεφαλής ε, ναβάρχου που μας έδωσε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν την μετακίνηση, τη διακίνηση αυτών των ανθρώπων έχουν σαφείς σχέσεις και με την τρομοκρατία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, κυρίως στα πλαίσια μιας επιστολής, η οποία, ε, αποστολής, συγγνώμη, η οποία κατά κάποιο τρόπο ε, ε, έχει, παρουσιάζει πολλά συνεκτικά στοιχεία διαφορετικά και για την ασφάλεια και για την εξωτερική πολιτική. Επίσης, μια έκκληση προς το Κοινοβούλιο για την ανάγκη συντονισμού, πώς να το πω, έτσι ώστε πραγματικά ε, να ε, συντονίζονται οι εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, δηλαδή από τη μία να βλέπουμε το προσφυγικό, από την άλλη όμως να βλέπουμε και να συντονίζουμε τις δραστηριότητες για την τρομοκρατία ε, και τις δραστηριότητες της εξωτερικής πολιτικής και όχι μονάχα ε, διαπραγματεύσεις στη Συρία, στην ε, Λιβύη και τα λοιπά, αλλά και για την εγκατάσταση της κυβέρνησης στην Λιβύη, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε τι κάνει ακριβώς και η UNAFOR MED, η οποία και αυτή παίζει το ρόλο της στα θέματα αυτά. Ε, γιατί είναι πολύ σημαντική η επιχείρηση και στις, ε, στα λιβικά ύδατα ε, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η διακίνηση ατόμων και να καταστρέφονται οι βάρκες των διακινητών. Ε, επίσης, Για να ξεκινήσει η δεύτερη και η τρίτη φάση αναμένονται οι δύο συμπληρωματικές ε, εντολές. Και Είδαμε ότι και από πλευρά των Ηνωμένων Εθνών είναι θετική ε, η άποψη όσον αφορά τη δεύτερη και την τρίτη φάση και η ίδια ε, η κυβέρνηση της Λιβύης θα πρέπει και εκείνη ε, να δώσει την επιβεβαίωσή της έτσι ώστε να γίνουν τελειωτικές οι δραστηριότητες αυτής της ε, αποστολής. Ε, είδαμε και πώς οι διακινητές αλλάζουν ε, τις στρατηγικές τους ακριβώς προσπαθώντας να αντιδράσουν στην αποτελεσματικότητα της αποστολής. Ε, και είχαμε και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ε, ε, αντιμετωπίζοντας από τους διακινητές υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο μάχες με τους διακινητές με τους οποίους είχαν έρθει με τοπικά ας πούμε αντίθετοι. Εν πάση περιπτώσει οι διακινητές αλλάζουν τρόπο δράσης λόγω της παρουσίας αλλά και της δράσης της αποστολής αυτής, πέρα δηλαδή από τη διάσωση των ζώων. Επίσης, τη δεύτερη μέρα είπαμε ότι μιλήσαμε και με τον ε, επικεφαλής ε, Ναύαρχο για τον τρόπο με τον οποίο ε, η αποστολή προσπαθεί να καλύψει και τη νέα διαδρομή, αυτήν την ανατολική ε, ε, αποστολή και ακριβώς όταν είμαστε εκεί μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης ε, λάβαμε γνώση της απόφασης σχετικά με το ΝΑΤΟ. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία ε, μια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο αποτελεσματική και να εφαρμόσει επομένως αυτή την διτή εντολή διάσωσης ζώων ε, και ε, αποκαθήλωσης ας πούμε όλου αυτού του συστήματος διακίνησης με πιο διευρυμένες διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει. Τώρα είναι παρόν και το ΝΑΤΟ. Ε, βεβαίως ε, η αρχή, η ιδέα ήταν ε, η Τουρκία και η, Ευρωπαϊκή, συγγνώμη, η Ελλάδα να βρεθούν και να συζητήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο να μην είναι αυστηρά και μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί παρισύφρισε το, το ΝΑΤΟ. Εμείς θα, είχαμε, θα προτιμούσαμε η συζήτηση να γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. εν πάση περιπτώσει ε, απ' την άλλη πλευρά βεβαίως και αυτό είναι μεγάλο θέμα συζήτησης. Ε, ε, το ζήτημα είναι οι πρόσφυγες εάν τελικά θα αποβιβάζονται σε ελληνικό έδαφος ή σε τουρκικό έδαφος σε περίπτωση δηλαδή που οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ τους σταματήσουν. Εν πάση περιπτώσει εμείς συνεχίζουμε ε, να δουλεύουμε για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τα εσωτερικά, ε, τις ε, ελευθερίες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Δουλεύουμε και τα εξωτερικά ζητήματα τέτοιων αποστολών, γιατί είπαμε ότι η αποστολή αυτή έχει την διπλή αυτή εστίαση ε, και τα εξωτερικά ζητήματα τα μελετούμε εδώ στην Επιτροπή ε, ΣΕΔΕ. Το σημαντικό είναι να στείλουμε ένα μήνυμα προς τους πολίτες της Ευρώπης ότι δηλαδή είμαστε σε θέση, έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να διασυνδέουμε, να κάνουμε πιο συνεκτικές τις δράσεις μας και, στο, και από εσωτερική και από εξωτερική ε, άποψη και όσον αφορά ε, την προστασία των ε, προσφύγων και όσον αφορά αυτών που εισέρχονται αυτή τη στιγμή στο, στο έδαφος ενώ ταυτόχρονα να καταπολεμούμε την τρομοκρατία. Ε, γιατί είδαμε ότι ακριβώς, ε, ε, να μην λησμονούμε πάντως ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έκαναν τις μεγαλύτερες επιθέσεις ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Πρέπει να δούμε βεβαίως και την χρηματοδότηση του, της τρομοκρατίας και να δούμε και ποια είναι η θέση και η επίπτωση που μπορεί να έχει η Ευρώπη όσον αφορά αυτές τις ροές στη ρίζα του προβλήματος, στη Συρία κλπ. Δεν ξέρω τώρα εάν η κυρία Πρόεδρος ε, θέλει να κάνουμε κάποια πρόταση ή εάν εσείς με τους ε, Προέδρους της ε, ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων θέλετε να κάνετε κάποια πρόταση έτσι ώστε να, ε, γίνουμε και πιο, να γίνουν οι πολιτικές μας και πιο αποτελεσματικές αλλά και πιο προληπτικές κατά κάποιο τρόπο έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σύνθετα προβλήματα. Thank you, for Σας ευχαριστούμε <clears throat> πολύ κυρία Γιάλα για όλα αυτά που είπατε. Είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει αυτή η οριζόντια προσέγγιση ε, και εγώ θεωρώ ότι υπάρχει διασύνδεση ανάμεσα στην εσωτερική και την εξωτερική ασφάλεια και αυτό αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, να σας πω ότι και εμείς μπορέσαμε όλα αυτά να τα εντοπίσουμε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ε, του briefing. Μας ε, ενημέρωσαν ε, σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών Μας ενημέρωσαν από τη διεύθυνση που ασχολείται με τη μαφία στην Ιταλία. Επίσης μας ενημέρωσαν και για την ε, ε, θαλάσσια αποστολή που αναπτύσσεται στην Ιταλία. Πράγματι έχετε δίκιο και αυτό ε, θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. διότι σε αντίθεση με ότι έχουμε συζητήσει όλα αυτά είναι σε αντίθεση με αυτά που πιστεύουμε. Θέλω λοιπόν να προσθέσω ότι αυτές οι τρέχουσες επιχειρήσεις ε, βασίζονται στην Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διάσωση ζώων ε, που διατρέχουν κίνδυνο στη θάλασσα. Δηλαδή ε, πρέπει κανείς να σώζει ανθρώπους που βρίσκονται στη θάλασσα ε, άρα δηλαδή δεν υπάρχουν άμεσες επιπτώσεις ε, με την ε, παράνομη εμπορία ανθρώπων. Είναι απολύτως απαραίτητο η κυβέρνηση της Λιβύης να επιτρέψει να λειτουργεί η Uniformed της, στη Σόφια και επίσης να καταδιώκει και τους διακινητές. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να σώζει κανείς ζωές. Αλλά πρέπει να περιοριστεί και αυτό το φαινόμενο της ε, διάδοσης ε, των ε, κινήσεων των διακινητών μέσα από τη μαφία. Ο κύριος Ντανζόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σε σχέση με αυτά που είπατε, εγώ θα ήθελα να είχα ε, ακούσει κάποιες διευκρινήσεις ε, για το πόσο αποτελεσματική είναι η επιχείρηση αυτή. Γιατί επιχείρησης πρόκειται με στρατιωτικά μέσα η εντολή της επιχείρησης είχε πολύ πιο αποφασιστικά στοιχεία από άλλες αποστολές αντίστοιχες και αυτό ακριβώς γιατί ο στόχος δεν ήταν μόνο η διάσωση ζωών αλλά και χτύπημα στα δίκτυα των διακινητών. Πρέπει να σας πω όμως ότι εγώ προσωπικά από την αρχή και επιβεβαιώνεται η άποψή μου από τις μαρτυρίες πολλών επαγγελματιών και ναυτικών. Είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για το πόσο η επιχείρηση αυτή μπορεί να είναι αποκλεισματική ως ε, την συνέλαβα τουλάχιστον για να σώζει ζωές. Θα μου πείτε δεν είναι και λίγο. Ναι, αλλά δεν είναι ο στόχος, ο μόνος στόχος αυτός. Γιατί έχουμε το εξή πρόβλημα, τον εξή περιορισμό. Όλοι οι ναυτικοί έχουν ηθική υποχρέωση να ε, βοηθούν κάποιον στη θάλασσα. Όπου και αν είναι, είτε είναι πλήρωμα ενός εμπορικού είτε ενός στρατιωτικού πλοίου, μπορείτε να του ζητήσετε να πυροβολεί ό,τι κινείται. Όμως η πρώτη αποστολή που έχει, εάν δει ένα σκάφος γεμάτο με μετανάστες, είναι να τους βοηθήσει και αυτό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν αξιοθαύμαστη δουλειά. Αυτό το δεχόμαστε όλοι. Όμως υπάρχει και το σκέλος της καταστολής που είναι σίγουρα ε, πολύπλοκο, είναι μακρόπνο, βασίζεται ε, και ε, σε σημαντική εκπαίδευση και ενημέρωση. Αλλά μπορεί να γίνει και αυτό. Γιατί πολύ σωστά και εσείς είπατε ότι τα δίκτυα διακινητών στην αρχή κάπως θορυβήθηκαν από την επιχείρηση αυτή. Αλλά είναι πάρα πολύ εύκαμπτα και ευέλικτα και αντιδρούν, προσαρμόζονται. Κατάλαβαν πολύ καλά λοιπόν ότι ούτως ή άλλως αν δεν υπάρχει, μπλοκ, ε, δεν υπάρχει μπλόκο ε, στα, Λιβανέζικα, στα ε, λιμάνια της Λιβύης, τι θα κάνετε εκεί. Θα καταστρέψετε ένα σκάφος, ακόμη και αν έχετε την εντολή, αν έχει πάνω το ανθρώπου, θα το καταστρέψετε θα σώσετε τους ανθρώπους αυτούς εντός εισαγωγικών. Παραμένει το πρόβλημα λοιπόν. Άρα στρατιωτική επιχείρηση, ακόμα και αν έχει την την εντολή, δεν μπορεί να κάνει τίποτε παραπάνω από την διάσωση των μεταναστών που πνίγονται στη Μεσόγειο. Επαναλαμβάνω, αν δεν αποκλειστούν ε, τα λιμάνια της Λιβύης. Και πώς αντιμετωπίζετε αυτή η δυσκολία. Έχουμε και το Συμβούλιο Ασφαλείας ε, ε, με τη δική του τη δικαιοδοσία. Γενικά και συγκεκριμένα, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τους διακινητές. Νομίζω ότι ξέρω λίγο πολύ την απάντηση, αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς που είδατε τους επαγγελματίε πώς ε, βιώνουν αυτή την κατάσταση οι ίδιοι. Πρόεδρος, ευχαριστώ. πριν περάσουμε και σε άλλα θέματα, να ήθελα, να, θα ήθελα να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο ότι οποιοδήποτε πλέον και οποιοδήποτε ναυτικός, είτε του εμπορικού ναυτικού, είτε του πολεμικού ναυτικού, έχει ως πρώτη αποστολή και πρώτο καθήκον να σώζει ζωές. Υπάρχει κέντρο συντονισμού και μπορεί να δίνει πληροφορίες οποτεδήποτε και σε οποιονδήποτε από την περιοχή. Και μπορεί να εξασφαλίσει ότι θα συμμετέχει στις ε, έρευνες και στη διάσωση οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος. Πολύ σωστά τα είπατε. Και πολλές φορές έχουμε πει ότι αυτή η επιχείρηση διέπεται από τη σύμβαση Σόλας. Είναι εδώ και η κυρία Γκόμες συμμετείχε και αυτή στην αποστολή. Για να μας πει και η ίδια τη εντυπώσεις αποκόμισε. Κύριε Γκόμε, ναι, ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν από την ε, αρχή, αλλά δεν έχουμε το χάρισμα του να είμαστε πανταχού παρόντε τέλο πάντων. Ήμουν στην αποστολή, είχαμε επαφέ με στρατιωτικούς, πάρα πολύ χρήσιμε ανταλλαγές. Αλλά αυτή, αυτή η αντίφαση, αυτά τα όρια ε, ισχύουν που είπατε έχουμε μια επιχείρηση που δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αν δεν υπήρχε εντατική συνεργασία με το Μάρε Σεκούρο, την Ιταλική επιχείρηση, που γίνεται σε λιβικά χωρικά ύδατα, με βάση προηγούμενες συμφωνίες που είχε η Ιταλία με τη Λιβύη. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως με τη δική μας επιχείρηση. Μπορεί να γίνεται μόνο σε διεθνή ύδατα. Και πολύ συχνά, όπως είπε και η πρόεδρος, μας έλεγαν ότι τον τελευταίο χρόνο έσωσαν 9.000 ε, ζωές. Είναι εντυπωσιακό αυτό το νούμερο. Άρα πρόκειται για πολύ σημαντικό επίτευγμα ήδη της επιχείρησης. Αλλά σε ό,τι αφορά τον άλλο στόχο ε, του να περιορίσει αυτά τα δίκτυα και τις κινήσεις των διακινητών, εκεί ήταν περιορισμένα τα αποτελέσματα. Ο Χαβιέρ Νάρτ ρώτησε τα μέλη της ε, αποστολής και αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν ότι Παρά την αποτελεσματικότητα μέχρι τώρα στη μείωση των ροών, από τη Λιβύη κυρίως, με τον καλό καιρό σίγουρα θα αυξηθούν πάλι αυτές οι ροές, είναι αναμενόμενο. Οι διακινητές που είναι οργανωμένοι, είναι οργανωμένες επιχειρήσεις ουσιαστικά και στη Λιβύη και σε άλλες χώρες. Και εντός Ένωσης όμως με σχέση που έχουν με τη μαφία κτλ. Προσαρμόζονται πάρα πολύ ωραία στις νέες συνθήκες. Και βέβαια θα μπορέσουν αυτά τα σκάφη να τα φτάσουν στα όρια με τα εθνικά ε, χωρικά της Λιβύης ε, και στα όρια τους με τα διεθνίδατα και να δώσουν μετά το σήμα για να πάνε να τους σώσει αυτούς τους ανθρώπους μετά η διεθνής αποστολή. Δεν ξέρω αν μιλήσατε γι' αυτό, αλλά σίγουρα πρόκειται για πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, το 30% του ΑΕΠ της Λιβύης. Έτσι μας είπαν. Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία. Αρχικά τα πιο πολλά ήταν αλληλευτικά σκάφη, ε, βάρκες mostly Από την Αίγυπτο και από μια άλλη χώρα, την Τινησία, που συμμετέχουν στα δίκτυα αυτές οι δύο χώρες. Αλλά τώρα εισάγουν ε, φουσκωτά από την Κίνα. Μπορείτε να καταστρέψετε όσα θέλετε από αυτά, αλλά θα χαρούν πολλοί Κινέζοι γιατί θα στείλουν κι άλλα. Άρα, όλα αυτά αποκαλύπτουν τα όρια της επιχείρησης. Υπάρχει όμως και μια άλλη επιχείρηση όπου συνεργαζόμαστε με θαλάσσια μέσα. Κάποια στιγμή καλό θα ήταν τις νέες αρχές της Λιβύης, όταν και εφόσον βέβαια αναλάβουν τα καθήκοντά τους, θα είναι καλό να τους βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε άλλη δράση υπερβαίνει την απλή θαλάσσια ασφάλεια. Να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν, να εκπαιδευτούν οι δυνάμεις ασφαλείας, όχι στη θάλασσα, αλλά και στην ξηρά. Είναι σημαντική αυτή η αποστολή. Όπως και η προηγούμενη αποστολή της και στην Λιβύη ήταν σημαντική, αλλά έχουμε όρια, υπάρχουν περιορισμοί. Και δεν θα έχει κανένα νόημα αν δεν υπάρξει συντονισμός με άλλα μέσα της εσωτερικής στρατηγικής από τη γάμα δέλτα home. Προσωπικά φοβούμε ότι αυτά τα όρια θα τα δούμε και με την τελευταία ιδέα αυτή της κινητοποίησης του ΝΑΔΑ σε μια παρόμοια επιχείρηση στο Αιγαίο. Εκεί νομίζω θα είναι ακόμα πιο προφανή τα όρια, πιο περιορισμένα και πιο αντιπαραγωγική θα γίνει αυτή η επιχείρηση γιατί τα δίκτυα των διακοινών φυσικά θα προσαρμοστούν και είναι σαφή τα όρια. Αν δεν υπάρχει στρατηγική για την αντιμετώπιση, τη διαφορετική αντιμετώπιση των προσφύγων και των μεταναστών, δεν θα αλλάξει κάτι. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα αίτια. Γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη. πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε ε, αυτή τη δυνατότητα να βγάλουν λεφτά με αυτόν τον τρόπο οι διακινητές. Πρέπει να κόψουμε το κέρδος. Μόνο αν εγκαταστήσουμε σαφείς, ασφαλείς ε, τρόπους στην Ορδανία, Λίβανο, Τουρκία, αν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να ε, ετούνται άσυλο εκεί. ή μετά να έρχονται με ασφαλή τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην δίνουν δουλειά εντό αγωγικών στους διακινητέ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρέμβαση. Σίγουρα η Ιταλική επιχείρηση, το Mare Nostrum, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Είχε ξεκινήσει νωρίτερα και ήταν διαφορετικέ πολιτικές συνθήκε στη Λιβύη. οι πληροφορίες που συνελέγησαν στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης είναι πολύ σημαντικές και για τη Unifor Med Sofia. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, θέλατε κάτι να προσθέσετε? Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, άκουσα και αυτά που είπε η κυρία Άννα να, αλλά να, δούμε, να σας πω και ποια ήταν η εντύπωσή μας. Είναι γεγονός ότι συνειδητοποιήσαμε τα όρια, ε, γιατί ε, όντως ε, είχε ξεκινήσει η δεύτερη φάση της αποστολής, αλλά είχε φτάσει και στα όρια τέλος πάντων της εντολής και της τωρινής, αλλά βεβαίως και σε σχέση και με τα όσα περιμένει από την νέα κυβέρνηση της Λιβύης. Ε, η εντολή ήταν ή το ένα ή το άλλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα έχουμε και το ΝΑΤΟ και λαμβάνοντας υπόψη και το θέμα της Ρωσίας και της Κίνας δεν έχει, ε, και η θέση τους δεν έχει τελειώσει, ναι, ε, έχουμε παραμείνει στο ή το ένα ή το άλλο. Θα εξαρτηθεί από την μελλοντική κυβέρνηση κυβέρνηση της Λιβύης. Αλλά ίσως εγώ επειδή είμαι νέα σε αυτές τις αποστολές, αυτό που μου φάνηκε πολύ σημαντικό ήταν ότι 22 κράτη-μέλη συμμετέχουν ε, σε μια επιχείρηση σε ευρωπαϊκή θάλασσα, ας πούμε, σε ευρωπαϊκά ύδατα στην Μεσόγειο θάλασσα. Ε, και ότι έχουν δουλέψει και όσον αφορά ε, την συλλογή πληροφοριών ε, για να δουν ποιες είναι οι οδοί που ακολουθούν οι διακινητές. Είδαμε ε, τι είδους ας πούμε ε, βάρκες χρησιμοποιούν στην ανατολική ε, διαδρομή και στη δυτική. Είδαμε ότι στη δυτική διαδρομή έχουν συχνά αυτές τις λαστιχένιες βάρκες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, αλλά εν πάση περιπτώσει ανταλλαγή πληροφοριών βάσει των νέων στοιχείων και κατάλαβαν καλύτερα πώς λειτουργεί αυτή η φρικιαστική βιομηχανία. Ε, και αυτές στις 9.000 ζωές ε, που σώθηκαν ε, από αυτούς τους ανθρώπους ε, πήραν πληροφορίες. Συνέβαλαν οι άνθρωποι πολύ μεταξύ αυτών των διασωθέντων στην αύξηση του όγκου των πληροφοριών μέσω μαρτυριών για τους διακινητές από τους διακινηθέντες ακριβώς για να μάθουν ποιοι ακριβώς τους περιμένουν στην αντίπερα όχθη, στην ευρωπαϊκή όχθη κάποιοι τους περιμένουν. Ορισμένες ε, κλήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες και από πολύ συγκεκριμένες χώρες και επομένως ε, μία ε, προεργασία όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι πάρα πολύ σημαντική. Και έχει δίκιο βέβαια ο κύριος Ντονζόν όταν λέει αυτά που λέει όσον αφορά τη την καταστροφή των ε, ε, πλοίων και τα λοιπά και ότι έχουμε ας πούμε Μαυριτανούς που μαζικά χρησιμοποιούν ε, αλλιευτικά σκάφη και τέτοια και τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια αναπτυξιακής βοήθειας και συμφωνιών τα κτλ. Αλλά ότι υπάρχει τουλάχιστον η δυνατότητα να καταστραφεί το πιο ορατό φυσικό κατά κάποιο τρόπο στοιχείο αυτής της ε, διαδικασίας την τρίτη μέρα, όταν ήρθαμε και συζητήσαμε ε, με τους συναδέλφους της αντίστοιχης Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας της Ιταλικής Βουλής, ε, υπήρξαν και ερωτήσεις σχετικά με την χρησιμοποίηση, την θεσμοθέτηση μάλλον ανθρωπιστικών διαδρόμων και αυτό ρωτήσαμε και τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης, με ποιο τρόπο αυτή η αποστολή θα μπορούσε να διασφαλίσει ένα τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, ε, αποκαθιλωθεί αυτή η βιομηχανία μέσα από, την, από τον καθορισμό ασφαλών ανθρωπιστικών διόδων. Και κάτι άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον, μας επιβεβαίωσαν ότι σε καμία στιγμή πέρα από την ε, κατάσταση ε, στην ε, Συρία και σε καμία στιγμή δεν σταμάτησε η μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και ότι η Κεντρική Τράπεζα σε καμία στιγμή δεν σταμάτησε να εργάζεται. Επομένως, πέρα από την όλη μπερδεμένη ας πούμε κατάσταση, η οικονομική διαδικασία συνέχισε να λειτουργεί ε, έτσι ώστε οποτεδήποτε ε, κληθούν να συνεργαστούν, να συζητήσουν οι διάφορες ομάδες, ε, θα έχει τη δυνατότητα η οικονομία της Λιβύης να ξαναρχίσει αμέσως ή, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε πολύ μικρό λογικό χρονικό διάστημα, εύλογο εάν λάβει κανείς υπόψη την περιπλοκότητα της κατάστασης. Uh, πριν λοιπόν κλείσουμε αυτό το σκέλος, το, το κομμάτι της συνεδρίασής μας, θέλω να προσθέσω ότι η Ιταλική εμπειρία από την αντιμετώπιση της μαφίας ήταν πάρα πολύ σημαντική για να αξιολογήσουμε την ενημέρωση που μας δόθηκε για την καταπολέμηση των μορφών και μοντέλων διακίνησης παράνομης διακίνησης ανθρώπων από τη Λιβύη προς άλλες χώρες της περιοχής. Προφανώς υπάρχει νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικέ ενέργειες και προφανώς υπάρχει και παράνομη διακίνηση μεταναστών στην Ευρώπη. Κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέρθηκε προηγουμένως είναι ο μηχανισμός SHADE που βασίζεται σε άλλα προηγούμενα επιχειρήσια. Τα λάντα παραδείγματος χάρη κάτι που είχαμε τότε να ε, παρακολουθήσουμε όλα τα προηγούμενα έτη, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα, όπως σας είπα, για το μηχανισμό SHADE, που αφορούσε επίσης και στην ε, ε, αποστολή UNAFOR ε, MED στη Σόφια. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία με τρίτα μέρη με τους άμεσα εμπλεκόμενους, γιατί με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς πράγματι να περιορίσει την παράτυπη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Κύριε Ντανζάν, θέλετε να σχολιάσετε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λόγια να σε ευχαριστήσω για τις ε, πολύτιμες διευκρινήσεις ε, που δώσατε. Εγώ με μεγάλο σκεπτικισμό βλέπω ε, την ε, επιβίωση αυτής ε, της, ή τη μακροημέρευση μάλλον αυτής της αποστολής. Γιατί όπως είπατε χρειαζόμαστε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό πληροφοριών έτσι ώστε να δουλέψουμε για να δούμε από πού ξεκινάει, προς τα πού πηγαίνει, ξέπλυμα χρήματος, εγκληματικές οργανώσεις. Ε, βεβαίως εδώ δουλεύουν με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί ε, να συνεχιστεί βεβαίως. Αλλά το ναυτικό το στρατιωτικό σκέλος ε, δεν θα μακροημερεύσει εύκολα γιατί κοστίζει εξαιρετικά ακριβά οι νευτικές ε, δομές των χωρών μας ε, πιέζονται οικονομικά πάρα πολύ και δυσκολεύονται ε, σε, να δεσμευτούν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και επιχειρήσεις γιατί βεβαίως και οι κοινή γνώμη, οι Ευρωπαίοι πολίτες κάποια στιγμή θα ζητήσουν το λογαριασμό ε, όντως αυτή η αποστολή ε, ξεκίνησε εν θερμό ε, και τότε οι πολιτικοί μας ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν εν θερμό να στείλουν τις δυνάμεις αλλά ε, νομίζω ότι ναι μπορούν να συνεχιστούν ας πούμε αστυνομικές επιχειρήσεις από ιταλικής πλευράς ε, επί λιβικού εδάφους όταν και εφόσον ε, υπάρξει συνεργασία με την Λιβύη αλλά όχι με πλοία του πολεμικού ναυτικού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρησή σας και θα ήθελα εδώ να κλείσω ε, θα ήθελα ε, ε, να, κλείσω την συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.